Thank you very much, whoever hushed everybody. So good afternoon, uh, everybody. A very warm welcome to our uh, session of the Internal Market Committee. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Μέχρι τις 6.30 είναι ε, θα κρατήσει η συνεδρίασή μας. Αύριο θα δουλέψουμε και πρωί και απόγευμα. Αύριο το πρωί έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα θέματα, πολύ ενδιαφέροντα θέματα, συγγνώμη, ε, αλλά και το απόγευμα επίσης για τις ε, κρατικές προμήθειες, ε, αλλά και για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Λοιπόν, Σήμερα το απόγευμα θα ασχοληθούμε με τον εξυγχρονισμένο ε, κώδικα, τελωνιακό κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα όμως να κάνω κάποιες ανακτήριες παρατηρήσεις. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω τους συναδέλφους. Καταρχάς να πούμε δύο λόγια για το πρόγραμμα πριν υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες ε, ψηλοαλλαγές, μικροαλλαγές, για να είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι συγητές ε, θα είναι παρόντες. Γι' αυτό και αύριο το απόγευμα θα έχουμε την ε, παρουσίαση της κυρίας Βερνιό. Λοιπόν, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι με την ημερήσια διάταξη. Την θεωρούμε ότι την έχουμε εγκρίνει. Να σας ενημερώσω επίσης ότι όπως συμβαίνει συνήθως ε, η σημερινή μας συνεδρίαση είναι web streamed, δηλαδή μας ακούνε και στο διαδίκτυο και το ακροατήριό μας θα ήθελα να το καλωσορίσω. Θα μπορούμε, μπορείτε στο, στην, στον ιστότοπό μας να βρείτε όλα τα έγγραφα και να ακούσετε τη συνεδρίαση μέσω του διαδικτύου. Ξέρετε ότι είχαμε ε, πολλές συνεδριάσεις το μήνα που πέρασε και το αποτέλεσμα των συνεδριάσεων αυτών θα σας ε, κοινοποιηθεί. Επίσης, η ομάδα εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο, η οποία προεδρεύει ε, υπό τον κύριο Αρίας, θα παρουσιάσει, παρουσιάσει το έργο της αύριο συντάσσουμε ένα σχέδιο συμπερασμάτων, το οποίο συζητήθηκε στις 10 Ιουλίου και ούτως ή άλλως υπάρχουν τα σχόλια στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, αγγλικά στο website. Επίσης, κάναμε και μια επίσκεψη στην Κύπρο εν ώψη της Κυπριακής Προεδρίας και τα αποτελέσματα της ε, επίσκεψης αυτής θα βρείτε στο website. Επίσης ε, θα ήθελα να καλωσορίσω τα τρία άτομα τα οποία ε, ήρθαν στην γραμματεία μας να σηκωθούν λίγο, να τους ξερίσουμε, να τους γνωρίσουμε. Η κυρία από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Σίγουρα δεν είπα το όνομά σας σωστά, αλλά θα το καταφέρω κάποια στιγμή. Η κυρία Αλεξάνδρα Κοτογλίδου, κάπως, ελληνικό το όνομα ακούγεται, από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Ε, ήρθε στο κοινοβούλιο τώρα και ο κύριος Κρίσιαν Κόλικ, ο οποίος ήταν στην Αλία, Γενική Διεύθυνση Αλίας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ήρθατε και οι τρεις εδώ και θα απασχοληθείτε πλήρως στο κοινοβούλιο. Τώρα, Σήμερα το απόγευμα θα, δημοσιευθούν, θα δημοσιευτεί μία μελέτη, η απλούστευση και ο, χρησι... του ε, εξυγχρονισμός συγγνώμη, του φόρου προστιθεμένης αξίας και η ψηφιακή αγορά. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία είχαμε θίξει και εμείς όταν συζητούσαμε την ψηφιακή αγορά. Λοιπόν, στα πρακτικά, έχετε μάλλον μπροστά σα. τα πρακτικά της συνεδρίασης τη 9 η και 10 η Ιουλίου. Εάν η γραμματεία δεν πάρει σχόλιά σας μέχρι το τέλος της συνεδρίασης της σημερινή ή τη αυριανή, θα θεωρήσουμε ότι τα πρακτικά έχουν εγκριθεί. Περνάμε τώρα στην έκθεσή μας για τις τροπολογίες που έγιναν στον τελωνιακό κώδικα της Ένωσης. Πρόκειται για μια αναδιατύπωση του κανονισμού και η εσωτερική αγοράς, η Επιτροπή Συγγνώμη Εσωτερικής Αγοράς και η Επιτροπή ε, Εσωτερικών Υποθέσεων θα γνωμοδοτήσουν επίσης. Έχουμε και τους σκιώδεις ε, εισηγητές, την κυρία Σιλβάνα Ράπτη από τους σοσιαλιστές. Ο κύριος Σμιτ δεν είναι εδώ. Η εισηγήτρια κυρία Λεγκρίπη είναι βέβαια. Ο κύριος Μπίλενης είναι εδώ. Και κάποιος που θα μιλήσει από τους πράσινους. Έχουμε αρκετούς σκιώδεις ε, εισηγητές. Θα μιλήσουν και εκείνοι καταρχάς και μετά ε, όσοι άλλοι θέλουν το λόγο. Καταρχάς όμως θα μιλήσει η κυρία Λεγκρίπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε εδώ σήμερα για να εξετάσουμε από κοινού την έκθεση για τον τελωνιακό κώδικα της Ένωσης. Ε, να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της σύνταξης αυτού του σχεδίου κανονισμού σεβάστηκα τη διαθεσμική συμφωνία για την τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, όπως είπατε κυρία κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μια αναδιατύπωση. Επομένω, τρι, οι τροπολογίε έγιναν για συγκεκριμένα τμήματα του κειμένου. Ε, επίσης, ε, υπάρχουν, υπάρχει δυνατότητα να υποβάλουμε και άλλες τροπολογίες ε, για τις διατάξεις που παραμένουν ε, ως έχουν στην πρόταση την οποία μας παρουσιάζει η Κομισιόν, δηλαδή το άσπρο κείμενο του κειμένου, το άσπρο κομμάτι του κειμένου και ε, πρέπει να υπάρξει πολιτική συμφωνία ανάμεσα στις ομάδες για να αγγίξουμε αυτό το άσπρο κομμάτι. Και ούτως ή άλλως θα κοινοποιήσω την θέλησή μου στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο να ε, υποβάλω νέες τροπολογίες, όπως θεσμικά είμαι υποχρεωμένη η αναδιατύπωση του τελωνιακού κώδικα είναι απαραίτητη, διότι πρέπει να τροποποιήσουμε, πρέπει να εξυγχρονίσουμε την τελωνιακή νομοθεσία, διότι μέχρι στιγμή η τελωνιακή νομοθεσία στηρίζεται στον κώδικα του 1992. Από τότε έχουν γίνει πολλές ε, τεχνικές ε, αλλαγές, ε, υπάρχουν εξελίξεις κτλ. Επίσης, ένας συνάδελφος το Δεκέμβριο του 2011 συνεισέφερε επίσης το εξυγχρονισμό του Ελληνιακού Κώδικα. Γι' αυτό η, η Κομισιό αποφάσισε να τροποποιήσει τον κανονισμό 450 με ένα νέο κανονισμό, ο οποίος θα ε, σεβόταν αυτό τους τρεις στόχους που μας παρουσίασε η Κομισιόν στις 26 Απριλίου όταν είχε έρθει. Αυτοί οι τρεις στόχοι ποιοι είναι. Καταρχάς να, να, να αναβάλουμε την ε, ημερομηνία για την εφαρμογή ε, του τελωνιακού κώδικα που είχε προβλεφθεί για τις 24 Ιουνίου του 2013. Και αυτή η αναβολή είναι απαραίτητη διότι ο καινούριος ε, κανονισμός ο οποίος απαιτείται δεν θα εγκριθεί εγκαίρως λόγω ακριβώς των καθυστερήσεων που έχουν ε, λάβει χώρα σε κάποιες χώρες. Επίσης ε, θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας, ο δεύτερος στόχος, να λάβουμε υπόψη μας τις συνέπειες της συνθήκης συνθήκη Λισαβόνα. Ε, πράξεις ε, κατεξουσιοδότηση, πράξεις εφαρμοστικές κτλ. Και μετά έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας για τα θέματα ασφάλειας ε, των διαδικασιών, των ηλεκτρονικών διαδικασιών. Λοιπόν, η βέλτιστη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί μια ομοιόμορφη και σωστή εφαρμογή της τελωνιακής νομοθεσίας που στηρίζεται στον τελωνιακό κώδικα. Αυτή η ανάγκη σύγκλησης της ε, νομοθεσίας είναι απαραίτητη και για τα κράτη-μέλη αλλά και για τους ε, εμπορευομένους, για τους ενδιαφερομένους. Επομένως ε, πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιες βάσεις που να προωθήσουν τον ανταγωνισμό στην κοινότητα σε σωστές, σωστές βάσεις κυρίως. Αυτό ήθελα να κάνω έτσι ώστε στο μέλλον να έχουμε μια σύγχρονη τελωνιακή νομοθεσία ε, που να ε, ικανοποιεί και τις τελωνιακές αρχές αλλά και τους εμπορευομένους, τους ενδιαφερομένους μάλλον. Λοιπόν, θα ήθελα ε, καταρχάς να, να, διευκρινίσω ότι οι τροπολογίες προσπαθούν να, κατα, να λάβουν υπόψη μια συμβιβαστική άποψη, διότι θέλουμε να διατηρήσουμε και κάποιες εξαιρέσεις σε κάποιες νέες αρχές, διότι ήθελα να συντάξω μια ισορροπημένη έκθεση. Και αυτό εμφανίζεται αυτή η ισορροπία στο νέο άρθρο 6 το οποίο σας προτείνω. Από τις αρχές ε, που αρχίσαμε να ανταλλάσσουμε απόψεις σας είπα ότι ήθελα να αλλάξω λίγο την, ε, την εξαίρεση η οποία, την οποία προτείνει η Κομισιόν στο άρθρο 6 παράγραφος 3. Η, η παράγραφος αυτή για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι το ηλεκτρονικό υπόβαθρο, αν θέλετε, πρέπει να υπάρχει για όλες α, τις ανταλλαγές ανάμεσα στις α, τελωνιακές αρχές ή στους ενδιαφερομένους. Και αυτό έχει σαν στόχο να διατηρήσει την ασφάλεια στις ε, ε, μετακινήσεις ε, των εμπορευμάτων στην κοινότητά μας. Όμως, το κείμενο το οποίο προτείνει η Κομισιό για την εξαίρεση αυτή δεν είναι σωστό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι πολύ καλά πλαισιωμένη η εξαίρεση αυτή για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα και στα 27 κράτη-μέλη. Ο κίνδυνος μιας εξαίρεσης ε, πολύ γενικής αυτή τη στιγμή είναι δύσκολος ε, να εφαρμοστεί. Ε, έτσι, αν μείνει το κείμενο όσο έχει, θα δημιουργηθούν ε, διαδικασίες δύο ταχυτήτων. Διότι θα υπάρχουν και τα κράτη-μέλη τα οποία θα κάνουν ε, τις απαραίτητες επενδύσεις στα συστήματα πληροφορικής και τα κράτη τα οποία δεν θα κάνουν. Ε, επίσης, εάν ε, παραμείνει γενικό το κείμενο, θα έπρεπε να επαναλαμβάνονται κάθε φορά οι, οι εξαιρέσεις ε, και σε, στο χαρτί αλλά και ηλεκτρονικά. Κάτι το οποίο δεν είναι σωστό ούτως ή άλλως. Γι' αυτό θα, ήθελα ούτω ή άλλως οι εξαιρέσεις ε, να χορηγούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. η ιδέα να δοκιμάσουμε νέες ε, διαδικασίες πληροφορικής για τα δεδομένα θεωρώ ότι είναι καλή. Προφανώς θα βελτιώσει το ε, ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όμως θα ήθελα αυτές οι δοκιμές να αφορούν μόνο τα μη ουσιαστικά στοιχεία του κανονισμού. Να περιορίζουμε τις δοκιμάσεις αυτές και αυτό είχε συμβεί και στον εξυγχρονισμένο το ελληνιακό κώδικα στο προηγούμενο στάδιο. Τώρα δύο σημεία τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά και για μένα αλλά και για άλλους που είναι η, η του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Αυτή όλη η όλη διαδικασία έγκρισης θεωρώ ότι είναι πολύ δαπανηρή και αυτοί οι οποίοι έχουν επωφεληθεί από αυτό το καθεστώς, οικονομική οικονομικοί ε, δηλαδή, θα έπρεπε να επωφελούνται από, από κάποιες απλουστευμένες τελωνιακές διαδικασίες. Γι' αυτό προτείνω τροπολογίες που αφορούν ε, την αξιοποίηση αυτού του εγκεκριμένου, του καθεστώτος ε, του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα και αυτό θα πρέπει να εμφανιστεί στο βασικό κείμενο, δηλαδή η αξιοποίηση και η αναγνώριση ε, αυτού του καθεστώτος πρέπει να αναφέρεται στο βασικό κείμενο. Είναι οι τροπολογίες από 10 έως 13. Επίσης προτείνω και τροπολογίες για την δημιουργία απλουστεύσεων, πραγματικών απλουστεύσεων, για όσους ε, αποκτήσουν αυτό το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, κυρίως αναφορά την ελάφρυνση των ελέγχων σε ε, σημεία εσόδου και εξόδου. Λοιπόν, αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το καθεστώς του, του, εγκεκριμένου, του οικονομικού φορέα. Είναι ένα στοιχείο ε, αξιοπιστίας και ασφάλειας, αν θέλετε. Ε, γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το αξιοποιήσουμε σαν το περισσότερο έτσι ώστε οι ανταλλαγές μας το εσωτερικό της Ένωσης να είναι πιο ασφαλής, αλλά και να ε, ενθαρρύνουμε τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκτήσει αυτό το καθεστώς να το αποκτήσουν. Θα πρέπει να δούμε βέβαια πώς θα χορηγηθεί αυτό το καθεστώς και κυρίως όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις ιδιαιτερότητες αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης για τις ε, διεθνείς ε, ε, ε, υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα τελωνία, συγγνώμη, ούτως ή άλλως θα σεβαστούμε τις υποχρεώσεις μας και προφανώς η το καθεστώς του οικονομικού φορέα, του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, είναι ένα καθεστώς το οποίο δέχονται μεγαλύτεροι εταίροι μα Ακόμα και έχουμε υπογράψει τους τελευταίους μήνες ε, και με τις Ηνωμένε Πολιτείες μια συμφωνία, όπου ακριβώς ε, προβλέπεται και αυτή ε, η... και αυτό το καθεστώς. Λοιπόν, έχουμε διεθνείς συμφωνίες που φτάνουν τα 700 δισεκατομμύρια και βλέπουμε ακριβώς ότι η Ευρώπη προχωρεί στη συμφωνία με τα διεθνή τελωνία και υπήρχε μια συμφωνία πριν από τις ΗΠΑ με την Ιαπωνία, την Σουηδία, την Νορβηγία και τον Καναδά στο σύντομο, στο άμεσο μέλλον. Λοιπόν, στηριζόμαστε σε κάποιες βασικές αρχές. Θα τις, τις ανέφερα ή τις αυτές τις βασικές αρχές. Επίσης έχουμε τις πράξεις ε, εκτέλεσης ε, και τις ε, εφαρμοστικές πράξεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε. Επίσης θα ήθελα να σας προτείνω κάποιες αλλαγές εδώ πρότεινα κάποιες αρχές τις οποίες θεωρώ θεμελιώδεις να εμφανίζονται στην βασική, στο βασικό κείμενο το ίδιο και όχι στις ε, ε, πράξεις κατεξουσιοδότηση και θα σας αναφέρω εν συντομία αυτές, ε, ποιες είναι αυτές οι βασικές αρχές. Είναι ο κεντρικός εκτελονισμός, οι βασικές αρχές ε, για την χορήγηση του ε, καθεστώτος εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, τα κριτήρια που διέπουν την εφαρμογή της, της χώρας προέλευσης ή της, του καθεστώτος προτιμησιακής προέλευσης. Τελευταίο σημείο, ουσιαστικό σημείο το οποίο θα ήθελα να δείξω, ε, είναι οι, αλλαγές, οι ενδεχόμενες αλλαγές των λευκών τμήματων του κειμένου και επιφυλάσσομαι να προτείνω αυτές τις τροπολογίες. Μέσα στα πλαίσια της αναδιατύπωσης αγγίζουμε μόνο τα γκρίζα τμήματα. Αυτό λέει η Διαθεσμική Συμφωνία. Πιστεύω όμως ότι θα ήταν ενδιαφέρον να προβλέψουμε και κάποιες αλλαγές στις διατάξεις που δεν έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλαγή μέχρι στιγμής στα λευκά τμήματα. Αλλά χρειάζεται μια συμφωνία πολιτική για να γίνει κάτι τέτοιο. Θα μπορούσαμε παραδείγματος χάρη αυτές οι αλλαγές να αφορούν το καθεστώς της προσωρινής αποθήκευσης. Όσον αφορά την προσωρινή αποθήκευση, θα πρότεινα αν καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία βέβαια όλοι μας, θα είναι να καταργήσουμε το καθεστώς διαδικασίας για αυτή την προσωρινή αποθήκευση. Για πάρα, πολλές, για πάρα πολλούς φορείς του, των τελωνίων, αυτή η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται διαδικασία με όλες τις συνέπειες που κάτι τέτοιο προβλέπει, διότι η προσωρινή αποθήκευση είναι κάτι συγκεκριμένο. Εάν γίνει όμως μια διαδικασία, αυτό ε, επιβαρύνει τις υποχρεώσεις και για τις εθνικές τελωνιακές αρχές, αλλά και για τους οικονομικούς φορείς. Προφανώς αυτό ήταν ένα παράδειγμα, έτσι. Πριν ε, προτείνω οποιαδήποτε αλλαγή στα λευκά τμήματα της ε, πρότασης κανονισμού που μας υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρω πάρα πολύ καλά <clears throat> ότι είναι ευαίσθητα τα πράγματα και πρέπει να το συζητήσουμε στην Επιτροπή μας με τους ε, σκιώδεις συζητητές. Όλα αυτά είναι μέσα στα πλαίσια της καλής συνεργασίας που έχουμε από την αρχή που συζητάμε τον τελωνιακό κώδικα, να το συζητήσουμε μεταξύ μας και να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Εάν τώρα επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία με τους σκιώδους εισηγητές, τότε κύριε Πρόεδρε θα σας ε, προτείνω και κάποιες αλλαγές και για αυτά τα λευκά τμήματα. Μέσα στα πλαίσια βέβαια του σεβασμού των διαθεσμικών συμφωνιών. Επίσης, ε, Είμαι ανοιχτή σε οποιασδήποτε προτάσεις, ερωτήσεις ε, που θα ήθελα να θέσουν οι σκιώδεις ε, εισηγητές, αλλά και όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Αν θέλουν να κάνουμε κάποια ερώτηση, στη διάθεσή σας. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κείμενο αυτό να επιτευχθεί μια συμφωνία και εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προς όφελος της Τελωνιακής Ένωσης και προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε την δυνατότητα με τα κείμενα τα οποία μας προτείνονται σήμερα, με την αναδιατύπωση, να εφαρμόσουμε μια ευρωπαϊκή τελωνιακή πολιτική που να είναι φιλόδοξη, διότι η Τελωνιακή Ένωση είναι ένας κρίκος στην εμβάνθηση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει σύμφωνος όλους εδώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντεγκρίπ, κύριε Ντεγκρίπ για την τόσο σαφή εξήγηση. Νομίζω ότι εστιάσατε στα ουσιαστικά θέματα τα οποία ε, πρέπει να μας απασχολήσουν. Τώρα, για το θέμα των τμήματων του κειμένου που είναι εκτός αναδιατύπωσης. Ε, θα το συζητήσουμε. Πρέπει όμως να περάσουμε κάποιες, από κάποια στάδια για να δούμε αν όλοι συμφωνούν. Και αυτό, ε, εάν επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα σε εσά και τους Κιώδης, θα το προχωρήσουμε. Τώρα, θα... θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω την ομάδα της Κομισιό ο κύριος Ζελίνσκι είναι ο επικεφαλής, είναι πολύ ισχυρή η ομάδα της Κομισιόν για να απαντήσει σε ερωτήσεις σας. Ο κύριος Ζελίνσκι ήταν και άλλες φορές εδώ και θα μας απαντήσει στα ερωτήματά σας. Λοιπόν, στον κατάλογο των ομιλητών έχω τους Κιώδες, ο κύριος Μάντερς, ο κύριος Σμιτ δεν είναι εδώ βέβαια. Κύριε Μάντερ, θα μιλήσετε για τον κύριο Σμιτ. Όχι. Καταρχάς η κυρία Ράπτη, κυρία Ρούλεν και ο κύριος Μπίλαν και μετά κύριος Βάρμα, Κανιέτη κτλ. κτλ. Αν θέλει και κανείς άλλος να ζητήσει το λόγο, που το λέτε. Καταρχάς η κυρία Ράπτη έχει το λόγο. Okay, right. okay. Mrs. Rapti, first. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πρώτα εσάς. Εύχομαι καλό χειμώνα γιατί είναι η πρώτη συνεδρίαση νομίζω που κάνουμε η δεύτερη, άρα έχω χάσει κάτι εγώ. Ε, εν πάση περιπτώσει, καλό χειμώνα, καλή δουλειά να έχουμε. Ε, το δεύτερο είναι να ευχαριστήσω την κυρία Λεγκρίπ, την εισηγήτρια. Και το τρίτο είναι να επισημάνω ότι καθόμαστε δίπλα-δίπλα και χρησιμοποιούμε και το ίδιο μικρόφωνο. Αυτά είναι δύο πολύ καλά σημάδια, εκτός από το ότι έχουμε μέχρι τώρα πολύ καλή συνεργασία. Έτσι λοιπόν, πολύ σύντομα, ε, σας λέω ότι έχουμε στην έκθεση αυτή να αντιμετωπίσουμε δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι το επί της ουσίας ζήτημα να λειτουργούν καλύτερα τα τελωνία. Το ζήτημα αυτό συνδέεται άμεσα με την πλήρη εναρμόνιση των διαδικασιών, αλλά και βέβαια με το χρόνο εφαρμογής των διατάξεων. Το δεύτερο θέμα είναι εξίσου σημαντικό, ίσως και περισσότερο από το πρώτο. Είναι η ορθή κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Μιλάω δηλαδή για την ισορροπία που χρειάζεται να πετύχουμε ανάμεσα στις πολιτικές αποφάσεις από τη μια και στη διοικητική αποτελεσματικότητα από την άλλη. Η κυρία Λεγκρίπ έχει καταφέρει μέχρι τώρα μία πολύ καλή ισορροπία και στα δύο προαναφερθέντα ζητήματα. Ε, για να έχει τώρα νόημα όλη αυτή η τεράστια προσπάθεια που γίνεται να αναθεωρηθεί ο ενωσιακός κώδικας. Θα πρέπει πραγματικά η εναρμόνιση των ηλεκτρονικών μέσων να είναι πλήρης. Εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει μια δύσκολη οικονομική συγκυρία ε, άρα προκύπτει ότι είναι μάλλον θεμητή η δυνατότητα προσωρινών παρεκκλήσεων, αλλά ασφαλώς με περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, ώστε να καταφέρουν τα κράτη-μέλη να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, να προσαρμόσουν τις υποδομές τους και κυρίως να εκπαιδεύσουν τους εμπλεκόμενους φορείς. Λέω ναι απερίφραστα στο να διευκολύνουμε τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς. Η κυρία Λεγκρίπ το παρουσίασε πάρα πολύ αναλυτικά το σημείο αυτό και ομολογώ, ε, θέλω να είμαι έτσι πάρα πολύ ειλικρινή στην κουβέντα που κάνουμε εδώ, ομολογώ ότι στην αρχή, στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε πριν το καλοκαίρι, ε, ε, ήμουνα λιγάκι επιφυλακτική, ήμουνα λιγάκι σφιγμένη πλην όμως α, ακούγοντας και την κυρία Λεγκρίπ με όλες τις λεπτομέρειες που δίνει. Ε, νομίζω ότι πρέπει να πούμε ναι στη διευκόλυνση των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Ε, βέβαια η συγγήτρια επισημαίνει πολύ σωστά ότι δεν είναι δυνατόν να αποφασίζονται τα βασικά κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για τη, οι φορείς για τη χορήγηση της σχετικής άδειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, μια και μιλάμε για τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς. Ε, θέλω να υπογραμμίσω πως δεν είναι, κατά τη δική μου γνώμη, δεν είναι δυνατόν ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας να μην βρίσκεται σε έδαφος της Ευρώπης, σε, σε ε, ε, έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, νομίζω ότι τίθεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα ασφάλειας από τη στιγμή που δεν έχουμε δυνατότητα ελέγχου. Επιπλέον, και πάντα έχοντας στο μυαλό μου, μένω πάντα στο θέμα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Έχω μία μικρή επιφύλαξη ε, στην τεκμηρίωση των κριτηρίων που προτείνει η κυρία Λεγκρή. Έτσι λοιπόν κρατώ λιγάκι αυτή την επιφύλαξη, ε, να γίνει και πιο ενδιαφέρον ο διάλογος και ε, θα καταθέσω ε, κάποιες τροπολογίες. Αυτό σκέφτομαι. Τέλος, συμφωνώ βασικά με τις περισσότερες προτάσεις που έχουν ε, αναλυθεί, που έχουν αναπτυχθεί για δύο ακόμη θέματα. Το ένα θέμα είναι η κατανομή των ελέγχων μεταξύ του τελωνίου αρχικής παραλαβής και του τελωνίου τελικής παραλαβής των προϊόντων. Και το δεύτερο ζήτημα είναι η απλοποίηση των κανόνων διασάφησης για την διευκόλυνση της ροής των εμπορευμάτων, αλλά, ε, το υπογραμμίζω, να τηρούνται όλοι οι απαραίτητοι κανόνες ασφάλειας. Ε, κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι ε, θέλω να είμαι αισιόδοξη ότι θα πάμε καλά, ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό ε, στο θέμα του ενωσιακού τελωνιακού κώδικα και εδώ απευθύνομαι όχι μόνο στην κυρία Λεγκρίπ που ηγείται αυτής της προσπάθειας που κάνουμε από την πλευρά του Κοινοβουλίου ε, απευθύνομαι και στην ομάδα της Επιτροπής που είναι πάρα πολύ δυνατή ε, και θυμάμαι και τις απόψεις που είχαν αναπτυχθεί την προηγούμενη πριν από το καλοκαίρι συνεδρίασης ε, και αυτό το λέω για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί αισθάνομαι ότι όλοι στην Ευρώπη, και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε συνομολογήσει, έχουμε παραδεχτεί, παρά τις επιμέρους διαφορές, ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να ξανανιώσει. Η εσωτερική αγορά είναι ε, η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να την τονώσουμε, πρέπει να την αναζωογονήσουμε. Και το θέμα του ενωσιακού τελωνιακού κώδικα είναι ένα πολύ πολύ σταθερό έδαφος μπορούμε εμείς να προσπαθήσουμε να το κάνουμε πολύ σταθερό έδαφος ώστε πραγματικά η εσωτερική αγορά να αναζωογονηθεί. Είναι κρίσιμο για τους Ευρωπαίους πολίτες για τους οποίους εργαζόμαστε και οι οποίοι μας έχουν εκλέξει και μας έχουν στείλει εμάς εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Uh, thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά κύριε Αράπτη. Ο κύριος Μάντας παρακαλώ, εξ ονόματος της ομάδας των φιλελευθέρων Άλντε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ζήτω συγγνώμη τον κύριο Σμιτ. Πολλά πράγματα αναφέρθηκαν. Έτσι λοιπόν δεν θα αναφερθώ στην εισαγωγή σε σχέση με αυτή την ενημέρωση. Ευχαριστεί ο κ. Σμιτ την εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι η ραχοκοκαλιά. Ένα από τα στοιχεία της ραχοκοκαλιάς είναι φυσικά για την δημιουργία της ενωσιακής ενιαίας αγοράς ο τελωνιακός κώδικας, ενωσιακός κώδικας και για τα εξωτερικά σύνορα και η απλούστευση του 2008 ήταν πολύ επικοδομητική και τώρα εργαζόμαστε με βάση μια πρόταση που έχουμε ενώπιόν μας <laughs> είναι υπέρ των ε, διαφοροποιήσεων αυτών. Συμφωνεί με την εισηγήτρια ότι όπως είχε συμφωνηθεί δεν θα πρέπει να αλλάξει κάτι. Κάποια κράτη-μέλη δεν μπορούν να ε, εγκρίνουν, να, να, κατανείμουν τα κονδύλια και γι' αυτό είναι υπέρ ο κύριος Σμιτ αυτής της συμφωνίας ε, και υπέρ της θα έλεγα μη υποχρεωτικής απαλλαγής θα θέλαμε να ξέρουμε ποιε είναι οι κατεξαίρεση περιπτώσει στο μέλλον. Αυτό είναι ερώτημα που θέτει ο κ. Σμιτ. Και κάποια ελαστικότητα για τι επιχειρήσει απαιτείται επίση για να καταστεί εφικτό ώστε οι συνδυασμένες αυτές διαφοροποιήσει να είναι δυνατόν να λειτουργήσουν θετικά στο μέλλον. Αυτά είχα να αναφέρω εξ ονόματο του κ. Όλε Σμιτ. Ευχαριστεί την εισηγήτρια και για την καλή συνεργασία και ευελπιστεί ότι θα συνεχιστεί η καλή συνεργασία στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ιδιαίτερα για το χρονοδιάγραμμα και για τις πτυχές του χρονοδιαγράμματος θα επανέλθουμε σε αυτά. Η κυρία Ρούιλε, σε σχέση με τον κύριο Μάντας, για τα φιλικά λόγια εξ ονόματος του κυρίου Σμιτ, συμφωνώ απόλυτα, ευχαριστώ και εγώ για την πολύ καλή συνεργασία. Ωστόσο πρέπει να ομολογήσω ότι δεν κατάφερα ακόμα να διαβάσω την έκθεσή σας η αγγλική μετάφραση κατά το μεσημερινό διάλειμμα έφτασε σε μένα και είχα ανηλυμένες υποχρεώσεις και δεν κατα... κατόρθωσα να την διαβάσω. Θα προσπαθήσω να το κάνω το δυνατόν ταχύτερα. Την έχω και στα γαλλικά ενώπιόν μου. Και φυσικά το ενδιαφέρον μου επικεντρώνεται όπως και του κυρίου Σμίτ για τι εξαιρέσεις. Και πρέπει να το πούμε, στην οικονομία υπάρχει στους οικονομικούς κύκλους μεγάλη ανησυχία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προ... ότι προτείνει πολλές εξαιρέσεις. Όλοι δεχόμαστε ότι υπάρχουν προβλήματα βέβαια και ότι οι προθεσμίες ε, και οι, προσδι... Ε, διορίες πρέπει να προσαρμοστούν και τη συζήτηση αυτή την είχαμε και σε σχέση με την έκθεση Σαλβίνη. Σαλβίνη βέβαια και είχαμε συμφωνήσει επ' αυτόν. Αλλά είναι σημαντικό και το χρονοδιάγραμμα, το δρομολόγιο να μην ε, παρακολουθεί και να μην παρεμποδιστεί, να μην δημιουργηθεί πίεση σε σχέση με τα κράτη-μέλη όσον αφορά τα συστήματα πληροφορικής και την ψηφιοποίηση και να καταφέρουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός επιτέλους. Διότι έχει κέρια σημασία για την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και την ευρωπαϊκή οικονομία να σημειωθεί ένα βήμα προς τα εμπρός. Να μην έχουμε πολλές εξαιρέσεις και τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να υλοποιήσουν το δρομολόγιο, το πρόγραμμα αυτό ε, στο χρονοδιάγραμμα όσο γίνεται καλύτερα. Συμφωνώ με αυτέ τι προτάσει για τις εξαιρέσει πρέπει να τις εξετάσω σε βάθο πιο εξειδικευμένα. Η πρόταση τη κυρία Λεγκρίπ είναι σωστή ότι αυτά τα κείμενα θα πρέπει να τα δούμε καταλεπτός ε, και να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις πτυχές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Ρούιλε. Από ό,τι κατάλαβα η γερμανική διερμηνία κάπως καθυστέρησε και γι' αυτό η γερμανική μετάφραση καθυστέρησε. Θα είναι όμως διαθέσιμη και νομίζω ότι ήδη θα είναι στη διάθεσή σας, έτσι. Εγώ έχω στα αγγλικά τη μετάφραση στη διάθεσή μου. Υπάρχει αγγλική μετάφραση, μια και την έχω εγώ στα χέρια μου. Νομίζω είναι διαθέσιμη η μετάφραση σε όλες τις γλώσσες. Καθυστέρησαν μόνο τα σλοβενικά και τα γερμανικά. Ναι, και εγώ τα είχα στα αγγλικά, αλλά με καθυστέρηση. Όλες οι γλώσσες θα είναι διαθέσιμες, δεν θα υπάρξει καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την κατανόηση, συνάδελφοι. Μπίλαν παρακαλώ. Ας ακούσουμε τις απόψεις σας ε, για την δική σας ομάδα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω σύντομα να αναφέρω αυτά τα στοιχεία που θέλω να τονίσω. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Ευχαριστώ για τις προσπάθειες που κατέβαλε να συντάξει την έκθεση με τον τρόπο αυτό. Και όσον αφορά τις, ε, ε, την έγκριση αυτών των διαδικασιών, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις τροπολογίες 9, 10, 11, 12, 13. Ευχαριστώ. Και θα προσπαθήσουμε να καταστήσουμε πιο θελκτικό αυτό το πλαίσιο για τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις. Ε, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια στα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται, όχι βέβαια αυθαίρετα, και γι' αυτό θα πρέπει οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να, λειτουργήσουν καλύτερα και να διευκολυνθούν. Και για τις ε, αντίστοιχες τροπολογίες για το άρθρο 181 είμαι κατά των πρόσθετων ε, βαρών που θα επομισθούν οι επιχειρήσεις. Θέλουμε πραγματικά να γίνει πιο ανταγωνιστική η Ένωσή μας. Ας αφήσουμε κάποιο περιθώριο, μεγαλύτερο περιθώριο για ελιγμούς, ε, για να κινηθούν ελεύθερα τα κράτη-μέλη. Και φυσικά υπάρχει και κάποια αναφορά στο άρθρο 106 του εξυγχρονισμένου τελωνιακού ε, κώδικα. Και πρέπει να δούμε ποιος θα έχει την ε, ε, έγκριση και θα δίνει τη σύμφωνη γνώμη για την απελευθέρωση αυτών των αγαθών. Σε σχέση με τις διαφορές που υπήρχαν όσον αφορά τις εθνικές νομοθεσίες για εισαγωγές και εξαγωγές. Όσον αφορά τις αντίστοιχε τροπολογίες για την εφαρμογή των κανόνων προέλευσης και όλους, όλες τις που αναφέρονται σε αυτά τα θέματα, 22 και 23 για παράδειγμα, δεν, δεν έχω βεβαιότητα αν αυτή η έκθεση, αυτό το πλαίσιο είναι το ενδεδειγμένο για τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Είχαμε θίξει αυτά τα θέματα, αλλά γνωρίζω ότι η Επιτροπή ε, Διεθνούς Εμπορίου είναι η αρμόδια εν τέλει για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγήτρια λοιπόν να τοποθετηθεί επί της σκέψης που βρίσκεται πίσω από την σύνταξη των τροπολογιών 78 ε, για παράδειγμα για την ε, διαγραφή της ε, υποχρέωσης να υπάρχει θηγατρική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί της. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπίλαν. Αυτά σε σχέση με τους πιο εισηγητές. Περνάμε τώρα στους ευρωβουλευτές. Ο κύριος Σουβάμπ, Νιέτη και Στάιλερ. Πρώτα ο κύριος Σουβάμπ λοιπόν. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Χαίρομαι φυσικά και εγώ που έχουμε αυτή την έκθεση που τη συζητούμε σήμερα. Παρότι και εγώ είχα την ίδια περίπτωση ότι ε, μόνο στα γαλλικά μπόρεσα να διαβάσω την έκθεση αυτή. Παρ' όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγητρία. Περιέχει σημαντικά στοιχεία που πρέπει όμως κατεπηγόντως να αλλάξουν, να τροποποιηθούν. Και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με την συνεργασία μας πρέπει να προχωρήσουμε. Γι' αυτό επτά σημεία πρόεδρε θα ήθελα να αναφέρω που θεωρώ ότι απαιτούν ένα εμβαθυμένο έλεγχο για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Διότι σε κάποια σημεία Πιστεύω ότι δεν έχει εξευρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ απογραφειοκρατικοποίησης και των αναγκαίων προσεγγίσεων για τις, ε, την δραστηριοποίηση των ε, εθνικών αρχών. Το πρώτο σημείο αφορά το 25 του σχεδίου έκθεσης. Αληθεύει με ότι δεν θέλουμε να έχουμε επιβαρύνσεις ε, σε σχέση με την έκθεση Le Grip. Όμως διευκολύνσεις αυθεντικές όσον αφορά τις ε, οικονομικές επιχειρήσεις ή τις άλλες επιχειρήσεις απουσιάζουν. Οι επιχειρήσεις πρέπει σε μεγάλο βαθμό να εργάζονται για να καταχωρούνται και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν αυτές οι διευκολύνσεις στον διοικητικό τομέα. Αυτό δεν είναι καλό, δεν διευκολύνει το εμπόριο, το βλάπτει μάλλον. Το δεύτερο αφορά πάλι το άρθρο 25. Εδώ όμως πρόκειται για τις κατεντολήν πράξεις, νομικές πράξεις. Για τους εμπλεκόμενους είναι σημαντικό να υπάρχουν ενιαίες διαδικασίες. Για παράδειγμα, αν θα υπάρχει, αν θα τίνει ευήκονους ε, μια δημόσια αρχή σε σχέση με το αίτημά τους. Αυτή η ενιαία νομική βάση θα πρέπει στην ίδια την έκθεση να κατοχυρώνεται και όχι να επαφήνεται στα κράτη-μέλη κατά το δοκούν ή κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Το τρίτο είναι το θέμα της ε, μη, προτι... Ε, της προτίμησης ε, όσον αφορά την προέλευση. Έχει εξαιρετική πρόταση η κυρία Λεγκρίπ που ανταποκρίνεται στο status quo και δεν αλλοιώνει τα πράγματα σε σχέση με το OCC. Παρόλα όλα αυτά θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσαμε λιγότερο γραφειοκρατικά και λιγότερο περίπλοκα να ε, αρθρώσουμε αυτό το πλαίσιο για να είναι πιο προσιτό. Το ε, τέταρτο αφορά την τελωνιακή αξία, τον καθορισμό της τελωνιακής αξίας και πόσο ε, ο, το, ο φόρος, ο δασμός ε, από τελωνιακής πλευράς καθορίζεται. Αυτό θα ήθε, γι' αυτό θα ήθελα και εγώ ίδιος να καταθέσω κάποιες τροπολογίες. Τα τρία επιπλέον σημεία μετά το 4 μέχρι το 7 μόνο προσωρινά ε, εντάχει θέλω να θίξω το, για το 18 όσον αφορά μια κατεντολήν πράξη το ίδιο αφορά και το άρθρο 182 και πάλι εδώ μια κατεντολήν πράξη που δεν είναι απόλυτα σαφής και για το 155 επίση. Αυτά τα οποία πιστεύω προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτά που η συνάδελφο Λεγκρίπ έχει καταθέσει ή έχει προετοιμάσει ως ε, τροπολογίες είναι θετικές ε, ε, συνέχειες αυτού του πλαισίου. Όμω, ποιε θα είναι, ποιες θα είναι οι εξουσίες τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσθέτω τη φωνή μου στην κυρία Ρούιλε, ώστε σε σχέση με τον τελωνιακό κώδικα να δούμε σε ποιο εύρος θα συμπεριληφθούν αυτές οι αρχές. Ευχαριστώ. Uh, thank ευχαριστώ πολύ. Κανιέτε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την Κωνσταντ, τη συνάδελφό μου, για την έκθεση που είναι πολύ λεπτομερής, εμπεριστατωμένη. Και τώρα περνάω στα Ιταλικά. Λοιπόν, πιστεύω όπως προτάθηκε από την κυρία Λεγκρίπ, η διευκόλυνση αυτών των τελωνιακών διαδικασιών είναι πολύ σημαντική για να καταφέρουμε να καταστήσουμε πιο λειτουργική και πιο αποτελεσματική την ε, εσωτερική αγορά και να μειώσουμε και τη γραφειοκρατική επιβάρυνση. Υποστηρίζουμε την πρότασή της ε, όσον αφορά το άρθρο 3 για την ανάγκη που υφίσταται τα κράτη-μέλη να μπορούν να ψηφιοποιήσουν ψηφιοποιήσουν τις τελωνιακές αυτές διαδικασίες στο μέτρο του εφικτού ώστε να μην υπάρχει ανάγκη γραπτό σε, έγγραφα, σε έντυπα να συμπληρώνονται διάφορα ε, τέτοια χαρτιά. Αυτό θα εξοικονομήσει και χαρτί και χρόνο και θα διευκολύνει τα πράγματα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, κατανοούμε ότι αυτό θα απαιτήσει δημόσιε επενδύσει. Ο προπολογισμό θα πρέπει να προβλέπει τα αναγκαία αυτά κονδύλια. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Όμω είμαστε διατεθειμένοι να επενδύσουμε σε αυτές τι δραστηριότητε γιατί θα βελτιωθεί το πλαίσιο για τις επιχειρήσεις μας και θα υπάρξει ένα γενικότερα εποφελές αποτέλεσμα, θετικό αποτέλεσμα για την οικονομία μας. Εκπλήσωμε κάπως πρέπει να πω ακούγοντας κάποιες φήμες ότι λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έπρεπε να αλλάξει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι θα έπρεπε να αφήνουμε όλες τις αποφάσεις ε, στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Απόλυτο λάθος αυτό, διότι με την συνθήκη Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δραστηριοποιηθεί και μάλιστα ενεργά σε σχέση με θέματα που αφορούν τελωνιακές διεργασίες και θέματα. Υποστηρίζω την κυρία Λεγκρίπ στη γνωμοδότησή της ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ροή αγαθών, τις ανταλλαγές αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να εξυγχρονίσουμε το σύστημα μεταφοράς αγαθών από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενεργά να συμμετάσχουμε στην ε, διαδικασία της έκθεσης αυτής. Έτσι λοιπόν ε, και από πλευράς μας θα υπάρξουν τροπολογίες. Και όπως και στο παρελθόν έγινε, Είμαστε βέβαιοι ότι από πλευρά τη κοινοβουλευτική μα επιτροπή η πρόταση που θα κατατεθεί θα είναι πολύ ισορροπημένη. Ισόρροπη προ ικανοποίηση και προ όφελο όλων για την ανάπτυξη τη ενιαία εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ και σε αυτό το γύρο. Τώρα τελευταία κυρία Στάιλερ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Το σημείο που ήθελα να αναφέρω αναφέρθηκε και, από, και προηγούμενα για την σπουδαιότητα της ψηφιοποίησης των τελωνιακών διεργασιών και την εξοικονόμηση που θα υπάρξει και υπάρχουν, και οι αναγκαίες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν, ωστόσο πρέπει να προχωρήσουμε και να καταφέρουμε με την ψηφιοποίηση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ε, να συγκλίνουμε ε, ε, στην προώθηση αυτών των θεμάτων και σε σχέση και με τις μεταφράσεις με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι υπάρχει τώρα διαθέσιμη και η αγγλική μετάφραση. Ευχαριστώ. Με ενημέρωσαν και μου είπαν ότι οι μεταφράσεις και στα γερμανικά και στα λετωνικά είναι και αυτές διαθέσιμες. λυπούμεθα για την ε, απουσία προηγούμενα και τώρα στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να εργαστούμε ώστε να καλύπτονται αυτά τα, αυτές οι ανάγκες. Ευχαριστώ. Αυτό το οποίο προτείνουμε να κάνουμε τώρα στη συνέχεια είναι να καλέσουμε τον κύριο Ζελίνσκι βρίσκεστε ακριβώς στην γραμμή προς τον κύριο Ζελίνσκι και τον αποκρύπτετε. Εσείς θα μπορούσατε λίγο να μετακινηθείτε. Λοιπόν, θα ζητούσα να μας σχολιάσετε κύριε Ζελίνσκι τα όσα ακούσατε μέχρι τώρα. Και θα ζητούσα μετά από την κυρία Λεγκρίπ να συνοψίσει για τις παρεμβάσεις των συναδέλφων και έτσι να δούμε και το χρονοδιάγραμμα και το τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια. Κύριε Ζελίνσκι, καλώς ήρθατε. Σας δίνουμε το λόγο. Παρακαλώ, με ιδιαίτερη χαρά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Εισηγήτρια, ήθελα να πω <clears throat> ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα με την έκθεση αυτή, είναι πάρα πολύ καλή. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά, το εκτιμούμε αυτό ιδιαίτερα. Τώρα, επί της ουσίας, σε γενικές γραμμές Υπάρχουν πολλές τροπολογίες με τις οποίες συμφωνούμε. Υπάρχουν τροπολογίες με τις οποίες, θα, τις οποίες μάλλον θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερο. Και υπάρχει και μια, ένας μικρός αριθμός τροπολογιών, τις οποίες θα θέλαμε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε με το Κοινοβούλιο ότι ενδεχόμενα δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στο κείμενο αλλά είμαστε ανοιχτοί για κάθε συζήτηση και να δοθούν ε, και από τις δύο πλευρές εξηγήσει. Λοιπόν, να σας πω ότι μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το σχέδιο ε, του κανονισμού. Θα κάνω πολύ σύντομες ε, παρατηρήσεις και για συγκεκριμένα σημεία, γιατί αλλιώς ε, θα σας κούραζα, θα μίλαγα όσο όλοι οι βουλευτές μαζί να σας πω ότι υπάρχει από πλευρά μας μια βασική ανησυχία. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση να υπάρχουν, να εμφανιστούν και να συμπεριληφθούν οι περισσότερες λεπτομέρειες στο βασικό κείμενο και όχι στα κείμενα τα οποία θα δημοσιευθούν εκ των υστέρων. Καταλαβαίνω βέβαια ότι ο βασικό στόχος είναι να ελεγχθεί η Κομισιόν. Αλλά και υπάρχει και μια τιμή γι' αυτό διότι και στις ε, πράξεις κατά εξουσιοδότηση υπάρχει έλεγχος. Και εάν στο βασικό κείμενο υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες, τότε θα γίνει άκαμπτο το κείμενο. Η κατάσταση αλλάζει. Στο παρελθόν ενδεχόμενα να μην υπήρχε δυνατότητα να διορθώσουμε εύκολα τα λάθη της Κομισιό. αλλά τέλος πάντων υπάρχουν αλλαγές. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα, αλλά αλλαγέ συμβαίνουν και στον εξωτερικό κόσμο. Και όταν υπάρχουν λεπτομέρειες στο βασικό κείμενο, τότε γίνονται. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα σχόλια που θα ήθελα να κάνω. Μετά, το δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω, ε, ίσως να μην είναι πολύ σημαντικό για να έχει πολύ μεγάλο βάρος, αλλά είναι σημαντικό για μας, είναι οι εξαιρέσεις. Καταλαβαίνουμε βέβαια πάρα πολύ καλά ότι οι εξαιρέσεις και τα κριτήρια θα πρέπει να καθοριστούν. Στα θέματα όμως προφορικής, το έχουμε συζητήσει με τα κράτη-μέλη και σε κάποια κράτη-μέλη δεν υπάρχει ε, δυνατότητα ε, εξέλιξης στην, ε, στην, στην πληροφορική ε, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένο στομέα τέτοιου είδους ε, εμπορίου ε, και δεν χρησιμοποιούν σε κάποια κρατημέλη κάποιες διαδικασίες που για άλλα κάποια κράτη είναι πολύ σημαντικές. Αυτή είναι μια εξήγηση. Στο θέμα των ΑΕΟ. Θέλω να σας πω ότι εδώ προσπαθούμε να καταλάβουμε καλύτερα και να δώσουμε στους δυνατόν περισσότερο ευκολίε. Ε, ε, περισσότερες ευκολίες. Και εδώ υπάρχει όμως ένα τίμημα το οποίο πρέπει να πληρώσουμε για τις διευκολύνσεις αυτές. Διότι εάν διευκολύνουμε υπερβολικά, τότε θα μας ζητήσουν να εισάγουμε όσο εδώ και περισσότερα κριτήρια διότι το εμπόριο διαφέρει, τα μέσα μεταφοράς, ο τρόπος μεταφοράς και εάν προσφέρουμε πολλές διευκολύνσεις θα πρέπει, θα μας ζητήσουν να εισάγουμε όλο ένα και περισσότερα κριτήρια. Και για να αποκτήσει κανείς ε, το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα θα είναι κάτι που θα γίνεται με μεγάλη δυσκολία και θα κοστίσει πάρα πολύ. Και, και αυτή δεν είναι η πρόθεσή μας. Αλλά τέλος πάντων εμείς προσπαθούμε να είμαστε στον πιο ευέλικτοι. Και μετά θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, όπως και σχόλια ε, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχόλια τα οποία πρέπει να αναλύσουμε και να τα κατανοήσουμε, διότι δεν είναι τα πάντα σαφή για μας τουλάχιστον. Αλλά είμαστε πάντα στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι και στο τέλος μάλλον της σύντομη παρέμβασής μου. Θα ήθελα να, ευχαριστήσω την κυρία Λουγκρίπ για άλλη μια φορά. Δεν θέλω να αλλάξω και τη γλώσσα, ε, τη γλώσσα μου κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, αλλά τέλος πάντων να ευχαριστήσω, Πρόεδρε, για την τόσο θερμή υποδοχή που επιφυλάξατε στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Ζελίνσκι λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι θίξατε κάποια θέματα ε, που συζητάμε και με, το Συμβου, και με το, την Κομισιόν αλλά και με το Συμβούλιο. Γι' αυτό είναι και τόσο ευαίσθητο το θέμα αυτό. Ε, προείδρευσα κάποιες, ε, κάποιους τριλόγους ε, πρόσφατα και ξέρω ότι το θέμα αυτό των εφαρμοστικών πράξεων, των κατεξουδότησης πράξεων είναι ένα θέμα που όχι μόνο εμάς αλλά και το Συμβούλιο ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ανησυχεί ιδιαίτερα. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο την κυρία Λεγκρίπη, για να σας απαντήσει και για να ε, κάνει και κάποια σχόλια του θέματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ σε όλες και όλες που μιλήσανε και εκφραστήκανε και φυσικά καταρχήν τους σκιώδης υπησίτες να ευχαριστήσω για τα διευκρινιστικά σχόλια. Διαπιστένω ότι υπάρχει μια ποικιλία όσον αφορά τις διάφορες πανεβάσεις είναι η πρώτη έκθεση που έχω την τιμή να σας παρουσιάσω. Είναι μια βάση εκκίνησης η οποία σίγουρα θα εμπλωτιστεί και σίγουρα θα συνεχίσει αυτό στην ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε. Λοιπόν, θα προσπαθήσω κατά κάποιο τρόπο να απαντήσω σε ορισμένες ερωτήσεις, ορισμένα από αυτά που ελέγχθησαν. Δεν έχω την πρόθεση ή τη δυνατότητα να απαντήσω σε όλα όσα ελέγχθησαν σε αυτό το στάδιο. Φυσικά λαμβάνω υπόψη τις ανησυχίες και το μεν και των δε όσον αφορά την αραμόνιση των ηλεκτρονικών συστημάτων, ότι εδώ πρέπει να διασφαλίσουμε κάποιες εγγυήσεις, τα θέματα των εξαιρέσεων και αυτά τα έχω εξάλλου προβλέψει σε μία επιστροπολογίες μου όσον αφορά τις εξαιρέσεις για τα συστήματα της πληροφορικής, για εξαιρετικές περιπτώσεις και ίσως θα πρέπει από την αρχή να ζητήσω συγγνώμη για τα προβλήματα μεταφραστικά που υπήρξαν, τα γλωσσικά. Ε, στα αγγλικά όμως υπήρξε από την αρχή μια διαθεσιμότητα. Τώρα, καταλαβαίνω επίσης, κατανοώ ότι γενικά στους βουλευτές που εξεφράσαν ότι υπάρχει μια επιθυμία να εδραιώσουμε εδώ κάτι, αλλά να διευκολύνουμε κιόλα τη διαδικασία και τα, το θέμα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Εξέφρασαν αυτό πάρα πολλοί συνάδελφοι εδώ. Σίγουρα πρέπει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να διευκρινίσουμε κάποια σημεία. Στις τροπολογίες που έχω καταθέσει που έχουν να κάνουν με θέματα προσδιορισμού αρμοδιοτήτων, θεσμικών οργάνων και εκτελεστικών οργάνων. Εγώ θέλησα πολλές φορές να διασφαλίσω κάποιες αρχές το βασικό κείμενο, για κάποιες αρχές δηλαδή που θεωρώ ότι είναι θεμελιώδεις. Μια προσπάθεια επαναδιάρθρωσης του κειμένου, του βασικού κειμένου, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούμε σαφέστατα τις λεπτομέρειες, ούτω ώστε η έκθεσή μου να μπορέσει να συμβάλλει τα μέγιστα. Εγώ θα επιθυμούσα να, να βρω κάποια ισορροπία όσον αφορά την ε, κατανομή των αρμοδιοτήτων και των, θα λέγαμε, εξουσιών ανάμεσα στα διάφορα θεσμικά όργανα. Δυστυχώ δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους. Ε, αναφέρθηκε Φερπίν το θέμα το θέμα εισαγωγή συγκεκριμένων οικονομικών φορέων στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Όντω υπάρχει ένα σημαντικό θέμα εδώ. Εδώ υπάρχει το θέμα της απαλλαγής ε, εξαιρέσεων, αλλά ειλικρινά υπάρχει εδώ θέμα διαλόγου για το δικαίωμα δηλαδή να έρθει κανείς στην Ευρωπαϊκή ή όχι επικράτεια. Είναι σίγουρα ένα θέμα το, για το οποίο θα συζητήσουμε πολύ ακόμα. Για πολύ. Αυτά ε, είναι λίγο σκορπισμένα αυτά, γενικά αυτά που ήθελα που μπορούν να σχολιάσουν σε αυτό το στάδιο. Σε γενικές γραμμές ευχαριστώ τους συναδέλφους. Σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να κάνουμε στην Επιτροπή μας και σίγουρα και με τα, συνεργασία με τα άλλα δύο θεσμικά όργανα. Έχουμε όμως χρόνο στη διάση μας να δώσω μια τώρα διευκρίνηση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των εργασιών μας τώρα. 16 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Ε, 16 Οκτωβρίου λοιπόν το μεσημέρι 12 στη συνέχεια ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί αρχές ε, Νοέμβρη 5-6 τώρα δεν έχει διασαφινιστεί ακριβώς η ημερομηνία σίγουρα θα έχουμε μια δεύτερη συνάντηση στην Επιτροπή για να δουλέψουμε μαζί Ενδεχομένω για συμβαστικέ τροπολογίες, ίσως γύρω στις 20 Νοεμβρίου και 29 Νοεμβρίου, κανονικά δηλαδή, θα πρέπει να ε, περάσει για ψηφοφορία το σχέδιο εκθέσεως και να δώσουμε εντολή. 29 Νοεμβρίου. Και στη συνέχεια οι εργασίες που θα μας οδηγήσουν ή μέχρι και τον την άνοιξη του 2013. Ευχαριστώ τους με και τους δε. Λαμβάνω υπόψη τις παρατηρήσεις, συγκριτική αν θέλετε, τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει και θα προσπαθήσω να ε, δώσω την κατάλληλη ε, αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Ευχαριστώ. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ηγείστε αυτού του τόσο περιπλόκου θέματος που χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Κυρία Λεγκρίπ, μήπως μπορείτε να με προσάξετε μισό λεπτό για το θέμα της παράτασης μάλλον της ε, διεύρυνσης ε, των αρμοδιοτήτων μας και για την αναθεώρηση ε, τμήματων του κειμένου που είναι εκτός της αναδιατύπωσης. Νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε, να το συζητήσετε εσείς μάλλον με τους συζητές πάρα πολύ σύντομα, διότι πρέπει να προβλέψουμε και τον χρόνο τον απαραίτητο για να γίνει αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει να συμφωνήσετε και με το Συμβούλιο. Τέλος πάντων, εσείς θα το αποφασίσετε, γιατί εσείς ηγείστε, αν θέλετε, του όλου θέματος, αλλά ε, πρέπει να ξεκινήσετε άμεσα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλου. πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ και περνάμε στο... στις ε, τροπολογίες του κυρίου Αρίας, μάλλον στις έκθεσεις του κυρίου Αρίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Είχαμε ένα κείμενο το οποίο μας ήρθε από την Κομισιό για να το μελετήσουμε, για να γίνει, για να γίνει συνεκτικός και αξιόπιστος ο τομέας της ψηφιακής ε, ενιαίας αγοράς. Έχουμε δύο συναδέλφους από την Κομισιό εδώ για να μιλήσουν, ξέρω του δύο θα το λόγο. Κύριε Αρίας, Δυστυχώς ο κύριος Αρίας είναι στο, ε, στο νοσοκομείο γιατί είχε πρόβλημα με τα γόνατά του. Τέλος πάντων, ο κύριος Σβάμπ θα είναι ο εισηγητής για σήμερα το απόγευμα, θα παίξει το ρόλο του εισηγητή. Και μετά η κυρία Ράπτη, που αντικαθιστά τον κύριο Κάμπος, ο κύριος Λούκε Γκάρντ, τον οποίο βλέπω εδώ, ο κύριος Άγκστρομ δεν είναι εδώ, δεν ξέρω αν θα έρθει και ο κύριος Μπίλαν αντικαθιστά την κυρία Μακλόφσκη. Βλέπουμε επομένως ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα ε, ατόμων που αντικαθιστούν ε, τους ε, σκιώδεις εισηγητής. Λοιπόν, έχουμε 110 τροπολογίες. 110 τροπολογίες. Ο κύριος Σβάμπ ξεκινάει. Ο κύριος Σβάμπ, ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πραγματικά σήμερα πρόκειται όπως είπε ο πρόεδρος ήδη για να έχουμε μια επισκόπηση για τις ε, τροπολογίες, τις πιο διαφορετικές τροπολογίες 110 και τώρα δυστυχώς βέβαια ο συνάδελφος Άριας δεν μπορεί να παραστεί σήμερα όμως παρόλα αυτά μπορώ να σας διασφαλίσω ότι η ε, εγχείρηση αυτή δεν θα είναι η αχίλια πτέρνα αυτής της έκθεσης με παρακάλεσε να ευχαριστήσω όλους όσους ε, κατέθεσαν τροπολογίες ο κύριος Άριας και πολλά από αυτά που κατατέθηκαν ως προτάσεις τροπολογιών εμπλουτίζουν το κείμενο της έκθεσής του, όπως αναγνωρίζει, και θα κάνει κάθε προσπάθεια τις καλές αυτές τροπολογίες, αυτές που θεωρεί θετικές, να τις ε, ε, δεχθεί για την προώθηση της ψηφιακής αυτής πτυχής ε, για την αγορά, για να μπορέσει να ενταχθεί στην έκθεσή του ε, το πλαίσιο αυτών των τροπολογιών. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα σκεπτικά, τις αιτιολογικές σκέψεις. Τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες ημέρες θα υποβάλει και συγκεκριμένες προτάσεις συμβιβαστικών τροπολογιών. Ίσως πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα για τα θέματα του ΦΠΑ, της πνευματικής ιδιοκτησίας, της ε, παράδοσης ε, και της προστασίας. Έχουμε διαφορετικές τροπολογίες που παρεκκλίνουν τόσο σημαντικά η μία από την άλλη που συμβιβασμοί δεν είναι εφικτοί παντού και δυσκολεύονται τα πράγματα. Τώρα σε σχέση με τις τροπολογίες για το ΦΠΑ, ιδιαίτερα τις τροπολογίες 54 έως 64, οι περισσότερες εκκινούν από το ότι εδώ κατεπηγόντως πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση, μια βελτίωση για την ψηφιακή αγορά διότι κατά τα άλλα τα εμπόδια των εσωτερικών νομοθετικών διατάξεων και των εσωτερικών νομοθεσιών θα εξακολουθήσουν να υφίστανται. Θα πρέπει να μπορέσει να δει ο εισηγητής τι μπορεί να επιλέξει από τα όσα έχουν προτείνει οι συνάδελφοι. Ε, μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατόν επιμέρους τροπολογίες πλήρως να προβλεφθούν ε, ε, όσον αφορά απόρριψη ή αποδοχή πρέπει να τις εξετάσει για τον εναρμονισμό των ε, διοικητικών δομών με θετικό πνεύμα την αντιμετωπίζει και το ενιαίο ποσοστό ΦΠΑ για τα ψηφιακά αυτά προϊόντα που ε, θέλει να τα εντάξει αυτά στην έκθεσή του ως προτάσεις. Το δεύτερο θεματολογικό πλέγμα αφορά την παράδοση, delivery, 54 64 τροπολογίες ή προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας από την άλλη πλευρά. Και οι δύο αυτές πτυχές θα πρέπει να συζητηθούν και να εξεταστούν σε μεγαλύτερο βάθος. Γι' αυτό μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν κάποιες προτάσεις συμβαστικών τροπολογιών ακόμα. Για το επόμενο θεματολογικό πλέγμα για την προστασία ε, δεδομένων και για την ε, γραμμή την οποία είχαμε υιοθετήσει μέχρι σήμερα, δηλαδή υψηλότερο βαθμό νομικής ασφάλειας και υψηλότερο βαθμό προστασίας δεδομένων, ώστε η ψηφιακή εσωτερική αγορά να μπορέσει να προαχθεί. Παρ' όλα αυτά όμως ο συνάδελφος Άριας λέει ότι αναγκαία ελαστικότητα πρέπει να διασφαλίζεται για τους παρόχους. Όμως με ένα συμβιβαστικό, με μια συμβαστική τροπολογία θα προσπαθήσει να καλύψει αυτό το τομέα. Προσωρινά θέλει να ευχαριστήσει όλους τους σκιώδους εισηγητές που κατέθεσαν τροπολογίε από τις κοινοβουλευτικέ του ομάδες και να εξετάσουν παρακαλεί αυτές τις τροπολογίε από τους άλλους ώστε να δούμε ποιε συμβαστικέ τροπολογίε μπορούν να επιτευχθούν. Ευχαριστώ. Well, thank ευχαριστούμε για αυτή την ε, σαφή παρουσίαση των απόψεων του κυρίου Άριας. Και να πω στου συναδέλφου ότι έχουμε τρει γνωμοδοτήσει από άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ και που θα θέλαμε να εξετάσουμε πλήρως μέσα σε αυτό το πλαίσιο και από την Πολιτισμική Επιτροπή και από την Επιτροπή Βιομηχανίας και από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που θα ψηφίσει σήμερα από ό,τι γνωρίζω ίσως θα θέλαμε να εξετάσουμε αυτές ε, τις ε, γνωμοδοτήσεις όταν θα έχουμε τη συζήτηση για τις τελικές συμβαστικές τροπολογίες. Σας ακούσουμε από τους σκιώδεις εισηγητές ή τους όσους εκπροσωπούν αυτούς. Η κυρία Ράπτη πρώτα, παρακαλώ. Μικρόφωνο παρακαλώ, μικρόφωνο. Merci. Alors, je Σχόλια του συναδέλφου Κάμπος για την έκθεση άρια. Οι τροπολογίες για αυτή την έκθεση γενικά είναι ισορροπημένες, ακολουθούν την ίδια γραμμή που επιβάλλει την αναγκαιότητα όσον αφορά ε, την ενιαία αγορά η οποία αξίζει μια καλύτερη λειτουργική, ένα καλύτερο λειτουργικό πλαίσιο αναγκαία όλα αυτά για την βιώσιμη ανάπτυξη η οποία αποβαίνει προ όφελο των καταναλωτών και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τα ταχυδρομεία και τα προβλήματα που έχουν να κάνουν μεταφορές σε, σε διασυνερικό επίπεδο, σημαντικό θέμα αυτό, προσπαθεί να ε, διασφαλίσει κανείς αυτό το χώρο, προβλέπονται κάποια μέτρα τα οποία δίνουν εγγυήσεις ούτως ώστε αυτές οι ε, παραδόσεις να γίνονται με σωστές τιμές και με το κατάλληλο τρόπο. Ένα ψηφιακό ενιαίο, μια ψηφιακή ενιαία αγορά θα πρέπει να προσφέρει μια πιο ευρεία προσφορά στον καταναλωτή με καλύτερες τιμές, αλλά φυσικά πρέπει να διασφαλιστεί ούτως ώστε ε, και αυτοί που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές να έχουν τη δυνατότητα προσέγγισης με σωστέ τιμέ. Ο κύριος Δεκάμπος θεωρεί ότι είναι αποφασίσει η να υπάρχει ε, πρόθεση αυτού του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά και με έναν τρόπο ο οποίος θα διασφαλίζει, θα δίνει εγγύησεις και δεν θα δημιουργεί προβλήματα την ενιαία ψηφική αγορά. Επίσης υπάρχει αναγκαιότητα ενός ελέγχου πολύ πιο αυστηρού από την πλευρά των θεσμικών οργάνων της Ευρώπης όσον αφορά τη μεταφορά, το, την υιοθέτηση των ιδιών από τις χώρες μέλη λαμβάνεται υπόψη ότι ένας κατακαιρματισμός δημιουργεί προβλήματα και ή μη σωστό τρόπο της ε, υιοθέτηση των ιδιών. Τα μέσα τώρα ε, ε, πληρωμών, με τα τηλέφωνα, τα κινητά, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δημιουργούν κάποια προβλήματα. Υπάρχουν τα θέματα κόστους, ε, διοικητικού κόστους που θα λέγαμε, που μπορεί να οδηγήσει σε κόστος πολύ καλύτερα από, την, από την υπηρεσία ή το προϊόν αυτό καθ' αυτό. Η δημιουργία νέων αγορών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης το θέμα χρηματοδότησης των καινοτόμων μικρών μεσαίων επιχειρήσεων μέσω προγραμμάτων που ήδη υπάρχουν ή με νέα προγράμματα θα πρέπει να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο το οποίο να οδηγήσει στην ένταξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ψηφιακή αγορά. Επίσης υπάρχει το θέμα των μη διακρίσεων, αναγκαιότητα αυστηρών κανόνων όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων και ανταλλαγή όσον αφορά το κέρδος ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Υπάρχει φυσικά και το θέμα των διενέξεων και πώς θα αντιμετωπιστούν. Θα πρέπει ο, ο καταναλωτής να έχει γνώση όλων αυτών των θεμάτων και θα πρέπει να διατυπωθούν με τον κατάλληλο τρόπο στις τροπολογίες. Εξ, εξ ονόματι του κύριου Ντεκάμπους, ε, σας ευχαριστώ. Thank you very much, Mrs. Rapti. Ε, Σας ευχαριστώ, κύριε Ρόκεγκαρτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης ε, τον εισηγητή, παρότι απουσιάζει βέβαια. Και εγώ διάβασα αυτές τις τροπολογίες με μεγάλο ενδιαφέρον. Φυσικά, όπως πάντα, έχουμε κάποιες διαφορές μεταξύ των ομάδων. Αλλά συνολικά πιστεύω ότι οι τροπολογίες αντανακλούν το γεγονός ότι ο κύριος Άριας πέτυχε μια σωστή ισορροπία σε σχέση με τα θέματα αυτής της έκθεσης. Σημαντικά βήματα πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ψηφιακή εσωτερική αγορά. Δεν θα μπορέσουμε όλα να τα κάνουμε ταυτόχρονα και διαμιάς. Όμως έχουμε τα θεμέλια, έχουμε τη διάγνωση των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν και αυτό είναι μια καλή εκκίνηση. Τώρα, σε σχέση με το έργο για τι συμβαστικέ τροπολογίε, θα ήθελα όμω να ολοκληρώσω από πλευρά μα, από πλευρά τη ομάδας Άλντε, λέγοντα ότι θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στι επιπτώσει για τι επιχειρήσει, πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα το κάνει εφικτό ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν αυτέ οι επιχειρήσει και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση που διατρέχουμε και διανύουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αυτό είναι σημαντικό στις διαπραγματεύσεις. Να δούμε, να επικεντρωθούμε το δυνατόν περισσότερο στις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ και προσβλέπω στις διαπραγματεύσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε, η κυρία Ρούλα αποσιάζει. Κύριε Μπίλε, εσείς εκπροσωπείτε Μακλάκεν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος ε, τη σκιώδους εισήγηση ε, Μακλάκιν θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με την έκθεση του κυρίου Άριας. Και εμεί υποστηρίζουμε το σχέδιο έκθεσης και την επικέντρωση στην ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης για το οποίο θέμα ο εισηγητή έκανε πολλά καλά πράγματα. Όμως κάποιες τροπολογίε υπάρχουν όπου η κυρία Μακλάκιν θέλει να επιστήσει την προσοχή σε αυτές ευελπιστώντας ότι θα μπορέσουν να ε, αναδιατυπωθούν σε συμβιβαστικές τροπολογίες. Η τροπολογία 27 αναφέρεται στα διάφορα συστήματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, copyright, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είναι ένα περίπλοκο σύνθετο θέμα. Είναι όμως εν δυνάμει ένας ε, μοχλός δημιουργίας ε, εισοδήματος. Τώρα, η επικέντρωση για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα θέματα είναι κάτι που συμπεριλαμβάνεται στην τροπολογία της 36. Σύμφωνα με το ψαχτήρι του Google, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ο μόνος τομέας που αυξάνεται και διευρύνεται αυτή τη στιγμή. Αν μπορούμε να θέσουμε σωστά θεμέλια στις υποδομές ώστε να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια και τα προσκόμματα όπως προτείνεται από την τροπολογία 41 υπάρχει τεράστιο δυναμικό. Συνδυάζεται με αυτά η ιδέα ότι η κατάρτιση για όλους ε, αυτούς τους εμπλεκόμενους θα πρέπει να προβλέπεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ένα πρόγραμμα το οποίο προβλέπεται και από την τροπολογία 40 που η κυρία Μακλάκιν ελπίζει ότι μπορείτε να υποστηρίξετε. Μια από τις ε, πρακτικές ιδέες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν για την προστασία των καταναλωτών είναι ένας θετικός ε, διοντολογικός κώδικας για όλες τις επιχειρήσεις, τροπολογία 85 από πλευράς της, ε, με ένα πολύ πιο καινοτόμο τρόπο για την αντιμετώπιση του ε, θέματος μιας κοινή ευρωπαϊκής ε, προσέγγισης. Μια κοινή τέτοια πρακτική θα μπορούσε να προωθήσει, να προαγάγει την εμπιστοσύνη, πράγμα το οποίο θα ήταν υποφελές. Και σε σχέση με τον εισηγητή έχουμε την τροπολογία 48 για παράδειγμα για να αντανακλάτε η άποψή της ότι υπάρχουν πολλά τεκμήρια όσον αφορά τον πίνακα επιδόσεων ε, scoreboard για να μπορέσουμε να ε, δραστηριοποιηθούμε ώστε να διευρυνθούν οι αναγκαίες αυτές οι υπηρεσίες. Όσον αφορά θέματα ΦΠΑ που διάφοροι ευρωβουλευτές προανέφεραν και σε σχέση με τις τροπολογίες τους, σε σχέση με την τροπολογία 62 η άποψη της κυρία είναι ότι πρέπει προσεκτικά να δράσουμε σε αυτόν τον τομέα και να επικεντρωθούμε στην απλούστευση των διεργασιών ΦΠΑ ώστε να αντιμετωπιστούν ε, οι επιβάρη, ε, τα γραφειοκρατικά βάρη των ε, επιχειρήσεων και να μην προωθήσουμε με δραματικό τρόπο μέτρα εναρμόνισης που δεν θα πετύχουν την ανάπτυξη που τόσο απεγνωσμένα χρειαζόμαστε σήμερα. Πρέπει να εξετάσουμε στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή τις αρμοδιότητές μας για αυτά τα θέματα και να μην θίξουμε, να μην ξεπεράσουμε τα εσκαμμένα και να μην αναμειχθούμε σε ε, αρμοδιότητες άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Επίσης, το σημαντικό θέμα της προστασίας των ανηλίκων θα πρέπει να διευρυνθεί όσον αφορά τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη. Γι' αυτό θα ζητούσε υποστήριξη για την τροπολογία της 99 από πλευρά σας. Άλλες τροπολογίες που υποστηρίζει η ΕΜΑ και, έχει, και που έχει καταθέσει προωθούν την ε, ε, προσέγγιση cloud computing ε, πράγμα το οποίο θα είναι επαναστατικού χαρακτήρα για τις δυνατότητες των επιχειρήσεων. Η σημασία όσον αφορά τα δεδομένα και την γνωστοποίηση και κοινοποίηση μέσα σε αυτό το πακέτο, έχοντας κάθε πολίτης δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε μια τέτοια σύνδεση η ΕΜΑ ΕΕ ζητήσει συγγνώμη για το ότι δεν ήταν σε θέση να παρακολουθήσει τη σημερινή συνεδρίαση, προσβλέπει όμως στη στενή συνεργασία με τον εισηγητή και τους άλλους κοιόδης εισηγητές, ώστε να εμβαθύνουμε σε αυτή την εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστώ. Uh, σε ευχαριστώ για αυτές τις ε, απόψεις που μας ε, μεταφέρατε και που δείχνουν το μεγάλο επίπεδο ενδιαφέροντος ε, που δημιουργεί αυτή η έκθεση. Και όπως αναφέρθηκε και από τον ε, κύριο Άριας, ε, υπάρχουν πολλές πτυχές που πρέπει να συμπεριληφθούν και να εμπλουτίσουν αυτή την προσέγγιση. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ ζήτησε τον λόγο. Άλλοι που θέλουν να παρέμβουν. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω οι 110 τροπολογίες πραγματικά αποδεικνύουν ότι υπάρχει θεμελιώδη συνένεση για την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών που είναι σημαντική υπόθεση για την ανάκαμψη της Ευρώπης και θα ήθελα κάποιες αποσαφηνήσεις από πλευράς της ΓΚΟΕ και από πλευράς ε, του Σουηδού συναδέλφου Γκούσταυσον που ζήτησε να διαγραφούν οι αιτιολογικές σκέψεις, για παράδειγμα το Α, που αφορά την τροπολογία 4 και την τροπολογία 13 η σημασία της ψηφιακής αγοράς που θα συνεισφέρει ώστε να γίνει πιο δημιουργική οικονομία και πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να διαγράψουμε αυτά τα εδάφια. Είναι δύσκολο να το κατανοήσει κανείς, ιδιαίτερα όταν ο συνάδελφος De Jong από την Ολλανδία είχε επισημάνει ότι εν τέλει αναγνωρίζουν και εκείνοι την αξία της εσωτερικής αγοράς για τη δημιουργία ανταγωνιστικών θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Θα ήθελα να μου, δοθούν, να επεξηγήσεις για αυτά τα θέματα. Δεν νομίζω ότι κάποιοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τέτοιες τροπολογίες. Κατά τα άλλα, ο σκιώδης εισηγητής από τις, ε, τους σοσιαλδημοκράτες νομίζω σε σχέση με αυτές τις ε, προσεγγίσεις, τουλάχιστον μεταξύ ΕΛΚ και Σοσιαλδημοκρατών μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι οι δοκιμασίες, οι δοκιμές ε, stress tests για το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σημαντική υπόθεση και από πλευρά του εισηγητού κυρίου Μίλαν που είχαμε ε, ψηφίσει την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συμπεριλάβει και την αναφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο στο πλαίσιο εκείνης της έκθεσης. Είναι νομίζω σημαντικό να έχουμε μία αναφορά και σε αυτό το πλαίσιο αυτής της γνωμοδότησης τώρα. Και το θέμα της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο είναι σημαντική υπόθεση και ελπίζω ότι θα υποστηριχθεί αυτή η προσέγγιση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Άλλος που θα ήθελε να λάβει τον λόγο και να παρέμβει για αυτές τις τροπολογίες για την ενιαία εσωτερική αγορά, τότε θα ζητούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Γενική Διεύθυνση Market να μας πούν δύο λόγια. Δεν ξέρω ποιος θα πει δύο λόγια για αυτά. Ο κύριος Τένοκ έχει τον λόγο λοιπόν για τα σχόλιά σας και τις σκέψεις σας για κάποιες από αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους όσοι είναι παρόντες εδώ και που υπέβαλαν τροπολογίες πάνω από 100, κάτι που δείχνει την σημασία της έκθεσης για τα θέματα επικοινωνίας. Τα καλά νέα είναι ότι η πλειοψηφία των τροπολογιών ε, μπορεί να γίνει δεκτή από την Κομισιό. Κάποιες, για κάποιες τροπολογίες έχουμε να κάνουμε κάποιες τεχνικές ε, παρατηρήσεις. Θα τις ε, υποβάλουμε και στην γραμματεία και στον εισηγητή διμερός. Αλλά σε γενικές γραμμές η, η, η, κατεύθυνση που ακολουθεί αυτή η Επιτροπή είναι η κατεύθυνση που ακολουθεί και η Κομισιό. Και, όπως είπε η κυρία το δυναμικό που παρουσιάζει, οι δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή ιστορική αγορά για την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας αναγκάζει να συγκλίνουμε τις προσεγγίσεις μας. Θα ήθελα να τονίσω καταρχάς ότι αυτή η ανακοίνωση υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 2012 και πάρα πολλά πράγματα έχουν ε, γίνει από τον Γενάρη και μετά είναι θέμα του τι κάνει η Κομισιό. Όχι μελλοντικά σχέδια έχει η Κομισιό. Αυτή τη στιγμή τι κάνει η Κομισιό και ε, αυτή τη στιγμή ε, ε παρακολουθούμε, ε, ακολουθούμε αν θέλετε αυτές τις εξελίξεις γίνεται η, η ενδιάμεση παρακολούθηση κάτι το οποίο ούτως ή άλλως κάνουμε ε, σε κάθε πρόγραμμα που εφαρμόζουμε, αλλά στις αρχές της επόμενης χρονιάς ούτως ή άλλως θα σας υποβάλουμε μία έκθεση ενημερωτική για τα όσα έχουμε πετύχει μέχρι τώρα στον τομέα αυτό. Υπάρχουν και δοκιμές αντοχής και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο για μας στην Κομισιό ε, είναι προ, προ, πρωτής Επίσης ε, υπάρχουν ε, και κάποιες ανησυχίες, θα γίνει και μια δημόσια ακρόαση για κάποια θέματα. Τέλος πάντων βλέπετε ότι ήδη εργαζόμαστε για την εφαρμογή της ανακοίνωσης. Ενώ ταυτόχρονα διαβάσαμε πάρα πολύ προσεκτικά τις τροπολογίες σας και θα, λάβουμε, θα τις λάβουμε υπόψη μας ως δόν περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε που μας δώσετε το λόγο. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Συμφωνούμε ούτως ή άλλως μαζί σας ότι θα πρέπει να παραμείνει πίεση, αν θέλετε, γι' αυτό όλο αυτό το, τη σειρά των μέτρων. θέλουμε να προχωρήσουν τα θέματα και θέλουμε κάποιοι από, αυτοί, αυτούς τους δείκτες να τους λάβουμε υπόψη μας και να εμφανιστούν στις εκθέσεις που αφορούν την ολοκλήρωση ενιαίας αγοράς. Γιατί θεωρούμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη οικονομική σημασία. Ο κύριος Γκούστασον θα πρέπει να σας απαντήσει ε, διμερός. Κύριε Σβάμπ, θέλετε να κάνετε κάποια καταρχητικά σχόλια εκ μέρους του κύριου Σβάμπ. Πρόεδρε, καταρχήν, εξ ονόματος του συναδέλφου Παύλου Αρίας, ναι. θέλω να ευχαριστήσω για τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις των συναδέλφων. Χαίρομαι φυσικά για το ότι προαναγγέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εργάζεται και επεξεργάζεται τα θέματα αυτά. Ειλικρινά όμως πιστεύω ότι όταν θα έρθει η ώρα να ψηφιστεί η έκθεση δεν θα εκπέσει διότι θα παραμείνουν επίκαιρα πολλά από αυτά τα θέματα που εμπεριέχει η έκθεση, ακόμα και αν επεξεργάζεται αυτά τα θέματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αξίζει αυτή η κοινή προσπάθεια και ο κύριος Άριας θα θέλει να συνεισφέρει από πλευράς του επ' αυτού του θέματος. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Right, well, um, we're going to have our next exchange views on the 10th of October. Θα έχουμε την επόμενη ανταλλαγή απόψεων στις 10 Οκτωβρίου. Θα υποβάλει και συμβαστικές τροπολογίες ο κύριος Άριας. Τότε θα δούμε <clears throat> τι λένε και τι αποστέλουν σε μας σε σχέση με τι γνωμοδοτήσει του ή άλλες κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Το χρονοδιάγραμμα είναι ότι θα ψηφίσουμε στις 11 Οκτωβρίου στην Επιτροπή Εσωτερική Αγοράς και θα έχουμε ψηφοφορία και τον Νοέμβριο και λαμβάνοντας υπόψη τι κοινοβουλευτικέ ομάδε που θα έπρεπε να συνεισφέρουν σε σχέση με τα θέματα αυτά. Προηγούμενα δεν είχε τύχει πλήρου συζήτηση η ψηφιακή αγορά και έτσι θα υπάρξουν και κάποια άλλα παράλληλα εγχειρήματα τα οποία εκτιλήσονται εκ παραλίλου και έτσι θα έχουμε μια μείζωνα συζήτηση νομίζω που αξίζει να διεξαχθεί από αυτόν και θα δούμε με τους συντονιστέ τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες για αυτά. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη στη συνέχεια είναι ψηφοφορία που είχε προβλεφθεί για τις 7 και 15. Δεν παρίστανται όλοι για αυτή την ψηφοφορία λοιπόν. Μια και τώρα είναι 16 και 30, θα έλεγα να κάνουμε ένα διάλειμμα για τσάι, για τσαγάκι, ώστε να υπάρξει χρόνος μετά από τις 6.30 μπορείτε αν θέλετε να πάρετε και καφέ, ένα μικρό σύντομο διάλειμμα για τσαγάκι και μετά θα ξανασυνέθουμε στις 17 και 15 ώστε να έχουμε το ψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που θα εξετάσουμε. Ευχαριστώ. Uh, uh, Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι όλοι σας. Θα περάσουμε σε σύντομη ψηφοφορία. Την προσοχή σας θα ήθελα για αυτό το θέμα παρακαλώ. Πρόκειται λοιπόν για μια ψηφοφορία που θα αντανακλά την άποψη αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για μια έκθεση από την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για από πλευρά του αρμόδιου εισηγητή. Λόγω του χρονοδιαγράμματος που είχε επιταχυνθεί από την, την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή δεν είχαμε χρόνο να διορίσουμε εισηγητή και να ακολουθήσουμε την κανονική διαδικασία. Ζήτησαν οι συντονιστές από τα μέλη των ομάδων τους να προετοιμάσουν κάποιες τροπολογίες. Δεν έχουμε επίσημη παρουσίαση εκτός από μέλη ομάδων που θέλουν να τοποθετηθούν για αυτές τις τροπολογίες 14 τροπολογίες συνολικά δεν ξέρω αν οι συντονιστές θέλουν ενεργά να παρουσιάσουν κάποιες απόψεις ο κύριος Σβάμπ είναι εδώ αν κάποιος από τους σοσιαλδημοκράτες θέλει κάτι να σχολιάσει ε, από πλευράς Γκρέφ που είχε καταβάλει προσπάθειες σε αυτό το θέμα και έχουμε και από άλλους συναδέλφους κάποιες τροπολογίες. Όσοι θέλουν να κάνουν κάποια σύντομα σχόλια προτού ψηφίσουμε, έχετε δικαίωμα να παρέμβετε. Ο κύριος Σβάμπ ζήτησε τον λόγο, θα παρέμβει πρώτος. Αν άλλοι θέλουν να παρέμβουν, θα μπορέσουμε να τους ακούσουμε, αλλιώς θα ψηφίσουμε. Σβάμπ, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον συνάδελφο Λούι Γκρέκ και την κυρία Τουρούνεν για την ε, ευμενή ε, τοποθέτηση να μπορέσουν να, δεχθούν κάποιες τροπολογίες ώστε να μπορέσουν και οι απόψεις του ΕΛΚ να αποκρισταλωθούν. <clears throat> Το ότι δεν είμαστε προηγούμενα έτοιμοι ήταν δική μας ε, ε, παράληψη. Ζητούμε συγνώμη. Και σε σχέση με άλλα θέματα που είχαμε δυσκολίες, τώρα όμως για αυτές τις τροπολογίες για τη θετική αντιμετώπιση θα μπορέσουν να, αντανακλούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ευρωπαϊκό εξάμεινο που άλλη διαδικασία θα έπρεπε να υιοθετήσουμε διότι το κεκτημένο της εσωτερικής αγοράς είναι ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση, όμως εδώ έχουμε μια κατεξαίρεση κατάσταση. Ευχαριστώ τον Λουι Γκρέκ και την κυρία Τουρούνεν. Ευχαριστώ. I mean, I agree with you. Συμφωνώ μαζί σας για τη διεργασία, με αυτά που είπατε. Καλύτερο θα ήταν να ακουστούν αυτές οι απόψεις από το να μην ακουστούν και εξ ονόματος των συντονιστών οι συντονιστές θα ήθελαν να διασφαλιστεί ότι κάποιες πτυχές για την ενιαία εσωτερική αγορά θα έπρεπε να συμπεριληφθούν όπως πρέπει σωστά στις πτυχές αυτού του εξαμήνου. Όμως μπορώ να πω ότι αύριο το απόγευμα οι συντονιστές θα συζητήσουν κάποιες προτάσεις, κάποιες τροπολογίες που προτάθηκαν για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε την ενιαία εσωτερική αγορά, την διάσταση, τη συνιστόσα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς πιο έντονα σε σχέση με το να είχαμε μια δεύτερη έκθεση που θα μπορούσαμε να έχουμε ένα συντονιστικό ρόλο εμείς ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή ώστε να μπορέσουμε συντονιστικά να δράσουμε για τα στοιχεία αυτού του εξαμήνου. Δεν θέλω να προδικάσω τη συζήτηση αυτή, αλλά ξέρετε ότι θέλουμε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε με κάποιες ευρύτερες συνιστώσεις για την συζήτηση που διεξάγεται ευρύτερα για αυτό το εξάμεινο. Άλλοι συνάδελφοι θέλουν να παρέμβουν. Ο κύριος Τζιον, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Η ομάδα μου δεν κατέθεσε κάποιες τροπολογίες για αυτή την έκθεση. Εγώ απλά θα ήθελα να εξηγήσω γιατί έχει συνέβη αυτό. Το πρόβλημα για την ενωτική ενωσιακή αριστερά είναι ότι είχαμε ένα πρόβλημα με το ευρωπαϊκό εξάμεινο ως θέμα Νομίζουμε ότι η καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και των ανισοτήτων είναι το πιο σημαντικό θέμα. Δεν έχουμε πρόβλημα με την ενιαία εσωτερική αγορά αφέ αυτής μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όμως είναι μια πολύ δυσχερής έκθεση για την ομάδα μας και έτσι δεν έχουμε καταθέσει κάποιες τροπολογίες. Θα καταψηφίσω αυτή την έκθεση ως έχει με την παρούσα της διατύπωση. Θα ήθελα όμως να επιστήσω την προσοχή στα μέλη της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής ότι επικεντρωνόμενοι στην ενιαία εσωτερική αγορά υπό το πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης δεν είναι κάτι που είμαστε εναντίον αφέ αυτού, απλώς αυτό ήθελα να εξηγήσω. Σίγουρα θα συνεισφέρετε στην περαιτέρω συζήτηση πώς μπορεί αυτή η συνιστόσα να ενισχυθεί περαιτέρω. Προσβλέπουμε σε αυτή τη συζήτηση λοιπόν μελλοντικά. Ας προχωρήσουμε με την ψήφιση δεν ζήτησα να, συγκεκριμένα να έχουν όλοι τις κάρτες τους. Νομίζω οι περισσότεροι θα τις έχουν. Αν μπορούμε να επιταχύνουμε τις διεργασίες θα μπορέσουμε έτσι να ψηφίσουμε. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν να ψηφίσουμε. Τροπολογία 4 της κυρίας Τούρουνεν με την προφορική τροποποίηση που έχει προταθεί. Όσοι είναι υπέρ κατά εγκρίθηκε με σαφέστατο τρόπο αυτή η τροπολογία. Τροπολογία 5 Τούρουνεν υπέρ κατά εγκρίθηκε και αυτή. Ε, δεν ζητώ να έχουμε τις αποχές, αποχές εκτός αν κάποιος θέλει υποχρεωτικά να ε, σημειωθεί. Η 6 του κυρίου Μάντερς υπέρ, κατά, σαφώς εγκρίθηκε. Η 7 του Ρούνεν υπέρ, κατά, σαφώς εγκρίθηκε. Η 8 του Ρούνεν υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Η 9 Γκρέκ υπέρ, κατά εγκρίθηκε. Η 10 γκρέκ υπέρ κατά εγκρίθηκε. Συμπεριλαμβάνεται φυσικά και η προφορική τροποποίηση που έχετε στον πίνακα. Η 11 γκρέκ υπέρ κατά εγκρίθηκε. Η 12 γκρέκ με την προφορική τροποποίηση υπέρ κατά εγκρίθηκε. Η 13 γκρέκ με την προφορική τροποποίηση υπέρ κατά εγκρίθηκε. Η 14 γκρέκ υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τώρα να πάρουμε τις ιδεολογικές σκέψεις 1 και 2 από κοινού. Ή έχουμε τις τροπολογίες 1 και 2 στα νέα σκεπτικά υπέρ, κατά και οι δύο εγκρίθηκαν. Τώρα, αιτιολογικές σκέψεις. Η τροπολογία 3 υπέρ, με την προφορική τροποποίηση υπέρ εγκρίθηκε. Λοιπόν, απλή υπόθεση ήταν, τελειώσαμε. Τώρα, ηλεκτρονική ψήφιση για να έχουμε τον αριθμό για την τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την τελική ψηφοφορία, για την τελική γνωμοδότηση προ έγκριση από την Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή. Άρχεται η ψηφοφορία. Άλλοι που, θέλετε να ψηφίσουν, που θέλουν να ψηφίσουν πέρα ψηφοφορία. 26 υπέρ λοιπόν, 27 υπέρ και ο κύριος Ντιόν ήταν κατά. Εντάξει λοιπόν, με, αυτή, με αυτό το αποτέλεσμα τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα διασφαλιστεί ότι αυτές οι τροπολογίες σε σχέση με την ψήφιση που έγιναν δεκτές θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκρέκα, Τούρουνεν και Μάντες που ανταποκρίθηκαν με αυτόν τον τρόπο την άλλη φορά θα έχουμε μια άλλη διαδικασία αυτό το θέμα τώρα ολοκληρώθηκε και έκλεισε Ζητώ λοιπόν όσοι θέλουν να φύγουν μετά την ψηφοφορία να αποχωρήσετε ήσυχα για να περάσουμε στο επόμενο σημείο, αν γίνεται. You're Do you want me to start now? Um, Κυρίες και κύριοι, προχωρούμε λοιπόν και περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι η συζήτηση για τη γνωμοδότηση για την πολιτική του ανταγωνισμού, για την έκθεση για την πολιτική του ανταγωνισμού, την ετήσια έκθεση που από την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα, την, είναι κύρια αρμόδια, Σάντσες Πρεσέντο, ο εισηγητής, συντάξης νομοδότησης για μας, ο κύριος Ανδρέας Σβάμπ. Πέντεργαστ, νομίζω εσείς είσαστε σκιώδης, ε, είσαστε η τελική σκιώδης εισηγήτρια γι' αυτό. Η κυρία Πρέντεγκας λοιπόν, εξ ονόματος του κυρίου Κοφεράτη. Ο κύριος Χατζημαρκάκης παρίσταται, τον καλωσορίζουμε, που θα είναι σκιώδης για την ομάδα της ΑΛΔΕ. Δεν βλέπω άλλους. Ο κύριος Μπίλαν για την ECR, ο κύριος Γιώμ για την ΚΟΕ, την Ενωτική Αριστερά. Έχουμε καλή παρουσία από τους σκιώδης εισηγητές, ασκιώδης ε, εισηγητές. Ξέρουμε ότι σε σχέση με την δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ο κύριος Σαλμούνιο, σε σχέση με τα θέματα που αφορούν την προστασία των καταναλωτών και τα θέματα αυτά είναι, ε, γνωρίζει ότι μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Καλωσορίζω τον κύριο Σβάπ και τον καλό να μας παρουσιάσει κάποια από τα θέματα που θα ήθελα να παρουσιάσει για την γνωμοδότησή του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ε, φιλική εισαγωγή. Κατά το παρελθόν, Άσλι Φόξ ήταν ε, ο συντάξης νομοδότηση για τη δική μα Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Ε, φέτος λοιπόν εγώ ε, διαδέχομαι την προηγούμενη αυτή σκιώδη ε, γνωμοδότηση για την ετήσια πολιτική για τον αγωνισμό που ετήσια παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τελευταία παρουσίαση ήταν για το 2010. Τώρα έχουμε για το 2011 τεσσαρακοστή ε, φορά που ε, υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι λοιπόν το Κοινοβούλιο όπως ζήτησε έχει αυτή την έκθεση και για αυτό το έτος ε, η έκθεση είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα αν επιτρέπετε να το πω, είναι πολύ πιο σύντομη η έκθεση και επικεντρώνεται στα ουσιοδέστερα σημεία που για τους ευρωβουλευτές και τους πολίτες έχουν το μέγιστο ενδιαφέρον. Αρχικά λοιπόν να πω ότι η τροποποίηση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δομή της έκθεσης καθιστά την έκθεση πολύ πιο ευανάγνωστη και πολύ πιο εύληπτη και αυτό είναι θετικό. Και πάντα έχουμε ουσιαστικά τα πιο σημαντικά στοιχεία που αναφέρονται σε σχέση με τον τύπο για τα θέματα ανταγωνισμού, ιδιαίτερα η ε, εξέταση όσον αφορά την περίπτωση Λίμπερο και το CDS όπου η Αρλίν Μακάθ, η πρώην ε, πρόεδρος αυτής της ε, Επιτροπής, υπό ειδική αρμοδιότητα για μια ειδική έκθεση είχε δραστηριοποιηθεί. Η ενιαία εσωτερική αγορά βρίσκεται πάνω-πάνω μέσα στο πλαίσιο του ενιαίου χώρου πληρωμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον χώρο πληρωμών είναι η Οικονομική Επιτροπή αρμόδια, αλλά έχουμε και την έκθεση Άριας που ε, προηγούμενα συζητήσαμε και τα θέματα που αφορούν την ηλεκτρονική κάλυψη του, των ηλεκτρονικών πτυχών του εμπορίου. Και εδώ έχουμε πάλι ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά θέματα ανταγωνισμού και ανταγωνιστικότητας και που απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια ισχυρότερη, πιο ενισχυμένη τυποποίηση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει ε, το θέμα του πριτανεύοντος ρόλου ή κυρίαρχου ρόλου ε, κάποιων παρόχων που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το χαιρετίζουμε και εμείς αυτό. Συνολικά είναι πολύ πιο σύντομη η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επικεντρώνεται σε κάποια σημαντικά θέματα. Ένα από αυτά είναι ένα από τα θέματα του, ε, των θεμάτων προστασίας των καταναλωτών. Έχουμε και θέματα όμως, ε, όπως προανέφερα, που αναφέρονται στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων που για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ε, συνδυάζονται και δίνουμε κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία ε, θέτει ο εισηγητής για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν κάποια από αυτά τα θέματα, όπως η επανακεφαλαιοποίηση των ευρωπαϊκών τραπεζών. Υπό το πλαίσιο της ενιαίας εσωτερικής αγοράς αυτό δεν είναι το ουσιοδέστερο. Ε, αν θα ενταχθεί όχι, αυτό μπορούμε να το δούμε στη συνέχεια τα θέματα αυτά έχουμε τις πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου που μέσα στο πλαίσιο δέσμης μέτρων ε, συνεισφέρουν όσον αφορά για παράδειγμα τους Δήμους, κοινότητες για το πώς μπορούν αυτές και αυτοί να εμπλακούν. Οι προτάσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτές τις επιδοτήσεις και το δίκαιο των ενισχύσεων έχουν τη σπουδαιότητά τους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απλούστευση για αυτό το πλαίσιο υποστήριξης προ, ε, επέλεξε να δώσει κίνητρα ε, με την παρακολούθηση των μέτρων αυτών ώστε να μην ε, υπάρχει η γραφειοκρατική επιβάρυνση στην οποία είχαμε καταλήξει στο παρελθόν. Όμως μια τέτοια αύξηση των επενδύσεων από το δημόσιο δεν θα πρέπει να παρακολεί την εξυγίανση των προϋπολογισμών και των δημοσιονομικών. Ιδιαίτερα αφορώνται εδώ οι υπηρεσίες νοσοκομείων, κλινικών, η κοινωνική στέγαση ε, και άλλου είδους τέτοιες παροχές που θα έχουμε υψηλότερα κατόφλια στο μέλλον ώστε να μπορέσουν μέσα στο πλαίσιο των ενισχύσεων και επιδοτήσεων να διαμορφωθούν πιο αποτελεσματικά. Είχαμε ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε κατά το παρελθόν και το οποίο εξακολουθεί να διαδραματίζει ένα ρόλο τώρα. Ο συνάδελφος Σάντσετ Πρεσέντο αναφέρεται στο roaming, στην περιαγωγή και στον τομέα τον ενεργειακό που πρέπει να τύχει περισσότερης προσοχής. Έτσι λοιπόν στο σχέδιο έκθεσης που συντάσσει η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς κάποια θέματα πρέπει να ενταχθούν επιπλέον. Πρόεδρε, οι αδρές γραμμές αυτού του πλαισίου έγκυνται στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μεριμνά να μην υπάρχει δεσπόζων ρόλος ή κυρίαρχη θέση κάποιων παρόχων στην αγορά ώστε να αποβαίνει προ όφελο των καταναλωτών ε, η προσπάθεια αυτή. Αυτά είναι τα ουσιοδέστερα από τα παραδείγματα που έδωσα. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτή την αρχή, με αυτή την προσέγγιση. Θα πρέπει μέχρι τις 8 Οκτωβρίου να καταφέρουμε να έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης που από πλευράς μου θα κατατεθεί στα μέλη, θα παρουσιαστεί στα μέλη της Επιτροπής μας, ώστε πριν από τα Χριστούγεννα να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Και γι' αυτό προσβλέπω σε όλα τα σχόλια των σκιωδών εισηγητών, αλλά και των άλλων υπόλοιπων συναδέλφων. Ευχαριστώ. Well, thank you. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις αρχικές σας παρατηρήσεις. Συμφωνώ μαζί σας. Πολλά υπάρχουν εδώ και είναι πολλά τα ενδιαφέροντα σημεία από πλευράς της έκθεσης ε, Sanchez Πρεσέντο. Και κάποιες από τις πτυχές αυτές που θέλουμε να συζητήσουμε και να εξετάσουμε, σίγουρο είμαι ότι οι συνάδελφοι θα παρέμβουν. Κυρία Πρέντεγκαστ, έχετε τον λόγο τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, μιλάω εξ ονόματος του Σέργιο Κοφεράτη ο οποίος λέει ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία που μας δίνεται τώρα για να δούμε την εσωτερική αγορά από μια γενική σκοπιά. Χρειάζεται βέβαια ε, πολλή δουλειά για να, είναι ανεξάρ... να υπάρχει μια ανεξάρτητη διάφανη αγορά που να σέβεται τα δικαιώματα των καταναλωτών. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία ανάμεσα στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ημών και των ομάδων καταναλωτών. Μέχρι στιγμής ε, δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται καμία κύρωση για την ε, παραβίαση των νομοθεσιών ε, για την, τον, τον ανταγωνισμό. Τα πρόστιμα εισπράττονται από τα κράτη-μέλη, ενώ εμείς, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν ταμεία με αυτά τα πρόστιμα για να καλυφθούν όλες οι διασυνοριακές δυσκολίες που δημιουργούνται οι συλλογικές αποζημιώσεις ε, και οι επανορθώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ο έλεγχος είναι πάρα πολύ σημαντικός ακόμα και για τους νέους τομείς δραστηριοτήτων μας. Ε, ας πούμε, ε, θα πρέπει να ενισχύονται οι διαδικασίες για τις ηλεκτρονικές πληρωμές πιστεύουμε ότι με τον κύριο Σβάμπ μπορούμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία έτσι ώστε να τελειοποιήσουμε την συνεισφορά της Επιτροπής μας. Και εδώ ολοκληρώνεται η παρέμβαση του κύριου Κοφεράτη. Ο κύριος Κατζημαρκάκης έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι ήρθε η χρονική στιγμή μετά από 20 χρόνια ενιαίας εσωτερικής αγοράς όχι μόνο ευγενικά λόγια να λέμε αλλά να θέσουμε το δάχτυλο επί του τύπου των ύλων. Η έκθεση επισημαίνει ότι η οικονομική κρίση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο με βραδείς ρυθμούς ε, μπορεί να ξεπεραστεί. Όμως δεν λέει με σαφήνεια και ξεκάθαρα η Επιτροπή ότι η ενιαία εσωτερική αγορά λειτουργεί, δεν λειτουργεί σωστά και αυτό έχει επιδεινώσει την κρίση περαιτέρω. Είναι απόλυτα σαφές λοιπόν ότι αν τα δει κανείς αυτά πιο προσεκτικά η απώλεια ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μειώθηκε. Αυξήθηκε η έλλειψη ανταγωνιστικότητας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση μέσα σε αυτά τα πλαίσια πολύ ρηχά, πολύ επιφανειακά αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζετε το θέμα των επιτοκίων που μετά από την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος φθηνό χρήμα ιδιαίτερα στις περιφέρειες και περιφερειακές περιοχές ε, συνεισέφερε και αυτό επιδίνωσε τα πράγματα ακόμα περαιτέρω. Αυτή η διασύνδεση παραγόντων δεν καθίσταται σαφής και εμεί ως Ευρωβουλευτές πρέπει να συμμετάσχουμε ώστε να αποσαφινιστούν αυτές οι διασυνδέσεις και οι αλληλουχίες με κάθε σαφή τρόπο ένα θετικό στοιχείο της ενιαίας εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να είναι ότι οι ισολογισμοί των κρατών μελών αυτής της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να ισοσκελίζονται. Χαιρετίζω το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε ένα μακροοικονομικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης κατά την άνοιξη του 2012, όπου οι διαφορές και οι ανισότητες των ισολογισμών φωτίζονται και διαφωτίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να, να, να μπορούμε να δούμε τις αρνητικές πτυχές Ελλάδα ή Ισπανία ή τις θετικές Λουξεμβούργο, Γερμανία. Όμω η Ευρωπαϊκή γερμανια ομως η ευρωπαικη επιτροπη δεν έχει κανένα μέσο ώστε να επιβάλλει κυρώσεις σε τέτοιου είδους παραβάσεις. Πρόκειται απλώς, απλώς για μια εικόνα, ένα στιγμιότυπο, μια φωτογραφία που έχουμε που αποτυπώνει την κατάσταση των πραγμάτων. Πρέπει όμως εμείς να δράσουμε αν θέλουμε η ενιαία εσωτερική αγορά να στεφτεί με επιτυχία και να μην είναι επιτυχία για κάποιους μόνο όπως συμβαίνει σήμερα και δεν είναι επιτυχία για όλους. Διαπιστώνουμε ότι μία ε, δημοσιοποίηση της ILO, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δείχνει την αύξηση ε, σε σχέση με την ανεργία. Έχουμε πάνω-πάνω Ναμίμπια και μετά Ισπανία-Ελλάδα που ακολουθούν με τη μεγαλύτερη ανεργία παγκόσμια παρακαλώ. Όλα αυτά μετά από 20 χρόνια ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίζει. Ζούμε ότι σε μια χώρα που παρουσιάζεται και αναφέρεται σε αυτή τη μελέτη έχουμε την τέταρτη μεγαλύτερη ύφεση παγκόσμια στην Ελλάδα το τέταρτο μεγαλύτερο υφεσιακό φαινόμενο στην ιστορία της. Και όλα αυτά μετά από 20 χρόνια ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Η αναποτελεσματικότητα των μέσων και εργαλείων μας είναι κάτι που πρέπει να καταστήσουμε σαφές. Διότι αυτά που αναφέρει η έκθεση, τα εργαλεία και μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, ψηφιακή ημερήσια διάταξη, ψηφιακό θεματολόγιο, διάταξη των ε, ε, δράσεων ε, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, όλα αυτά είναι χωρίς αποτέλεσμα όπως βλέπουμε. Γι' αυτό οι προσπάθειες του Ευρωκοινοβουλίου πρέπει να συνεχιστούν και παρακαλώ ο Πρόεδρος να δραστηριοποιηθεί ώστε με την κυρία Μπόλς να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί για την ε, Δημοσιονομική Ένωση. Fiscal Union. Έχουμε το Six Pack και το Two Pack, την ε, εξαπλή πρόταση και την ε, διπλή πρόταση. Υπήρξε τροχοπέδηση των πραγμάτων επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τελικά απο, απαγκιστρωθήκαμε και μπορέσαμε να κινητοποιήσουμε αυτά τα θέματα για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Η έκθεση αναφέρει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, την δυσλειτουργία των οίκων αξιολόγησης. Και μέχρι σήμερα σε σχέση με την αρνητική τους δράση για την ανταγωνιστικότητα δεν έχουν αναφερθεί πολλά πράγματα. Θέλω να το αναφέρω αυτό τυχαία εντό εισαγωγικών η Γαλλία, η Γαλλία υποβαθμίστηκε από την Standard Poor's και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπόρεσαν να διαπιστωθούν κάποιες παρατυπίες και κάποια ολιστήματα. Ας είμαστε όμως ειλικρινείς. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητήθηκε να δημιουργηθεί ένα σήκος αξιολόγησης, ένα ίδρυμα αξιολογήσεων ώστε να μπορούμε να δρούμε πιο έγκαιρα και ταχύτερα, διότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα για την Ευρώπη όσο βλέπει κανείς από αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χατζημαρκάκη. Ο κύριος Μπίλεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις εξ ονόματος του κυρίου Άσλι Φόξ που είναι ο ισχυώδης μας. Ένα ουσιαστικό στοιχείο για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς είναι μια συνεκτική πολιτική ανταγωνισμού, διότι και τον καταναλωτή βοηθάει αλλά και επιτρέπει τον, τον θεμητό ανταγωνισμό. Και η Κομισιόν προκάνει μια πρόταση που βοηθάει μόνο τον καταναλωτή, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, η σημασία των μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή την περίοδο της κρίσης και θα πρέπει να ενδυναμώσουμε την πολιτική ανταγωνισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ανοιχτές και ε, διάφανες αγορές. Αλλά οποιοδήποτε νέος κανονισμός δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα περίπλοκος, γιατί αυτό θα ε, θέσει σε κίνδυνο την ανταγωνιστική μας ε, θέση. Ε, θα πρέπει να έχουμε σαν στόχο μακροπρόθεσμους στόχους όπως η κοινωνική ευημερία, η υποστήριξη της ανάπτυξης, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ανάπτυξη και στη δομέα της έρευνας ο ανταγωνισμός είναι μια κινητήρια δύναμη και για παραγωγικότητα και, ε, πιο, και καλύτερη χρήση της τεχνολογίας και των πόρων. Ε, νομοθεσία για ε, κατά τον τραστ θα πρέπει να μας επιτρέψει έτσι ώστε να μην δημιουργούνται δεσπόζουσες θέσεις και να επιτρέπεται είσοδος μικρών φορέων. Οι μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις για μας είναι η βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και ο κύριος Ντιγιόγκ. και εδώ ολοκληρώνουμε τους σκιώδεις ηγητές των ομάδων και μετά αν θέλετε ε, συνεχίζουμε. Κύριε Ντεγιόγκ, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι στον ανταγωνισμό υπάρχουν ε, τρεις παράγοντες διαταραχής. Η κυβέρνηση, η, ε, η αλληλεπίδραση καταναλωτών και παραγωγής και η, η διαμάχη ανάμεσα σε επιχειρήσεις. Έχουμε με το δημιουργία στην εσωτερική αγορά συνθήκων για ανταγωνισμό χωρίς να εμποδίζεται το θέμα του ανταγωνισμού. Είναι σημαντικό να δούμε για, με συνεργασία με τους ε, καταναλωτές. Εγώ ήμουν σε ένα οδοντίατρο σήμερα το πρωί και αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι προσπάθησε να μου πει ότι προσπαθούσε να μου πει μια ενδιαφέρουσα τιμή μέσω τηλεφώνου. Η διατάξη όμως δεν ήταν πολύ σεφής και έτσι δεν το πέτυχε. Εγώ αυτό που επιθυμώ είναι μέσα σε αυτήν εδώ την έκθεση να, να συζητηθεί μια τέτοια ε, πτυχή. στι κάτω χώρες βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα φάρμακα φερπίν. Αυτό το βλέπω ανάμεσα στις χώρες. Έχουμε μια νέα αγορά. Τη στιγμή που έχουμε μια νέα αγορά, γιατί βλέπουμε κάτι τέτοιο. Γιατί το ίδιο φάρμακο είναι πολύ πιο φθηνά φερπίν σε μια χώρα σε σχέση με κάποια άλλη. Και επίσης να πω ότι υπάρχει μια συγκέντρωση θα λέγαμε που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, αυτό συγκεκριμένα στον χώρο των ε, μέσων μαζικής επικοινωνίας. Στα οπτικοακουστικά μέτρα, στο ίντερνετ, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι είναι μία συγκέντρωση τεράστια η έκταση αυτού του θέματος. Κάτι το οποίο έχει επιπτώσει ε, στον ανταγωνισμό. Κάτι το οποίο επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιθυμεί περισσότερο, περισσότερο ανταγωνισμό υπέρ του καταναλωτή. ε, Απ' τη μια έχουμε κάτι περιπτώσει όπω η General Motors Φερρυπή, όπου επειδή ήταν πολύ μεγάλη επιχείρηση, θεώθηκε ότι έπρεπε να την στηρίξει κανεί από την πτώχευση. Ε, στην Ευρώπη τώρα τι ακριβώ γίνεται, πώ έχουν οι κανόνε, δεν πρέπει να έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο ανταγωνισμού. Όσον αφορά τώρα τι σχέσει ανάμεσα στου καταναλωτέ, Φερρυπή είναι αυτό που βλέπουμε στην Ολλανδία. Ε, είναι ότι δεν έχουμε μια κατάσταση μορπολιακή, αλλά τι διαπιστώνουμε ότι φέρπιν η αλυσίδα Hain, σούπερ ε, που κάνει κάποιες φέρπιν ε, προσφορές με μια φέρπιν έκπτωση 2% κάτι το οποίο οδηγεί σε κάποιες άλλες ε, ε, επιδράσεις και πιέσεις φέρει πίν ε, αγρότες. Ευχαριστώ. Ναι. Κανεί Um... Κανείς άλλος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Εάν όχι θα ήθελα να κάνω εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Θα ήθελα να χαιρετήσω και την παρουσία της εκπροσώπου της Κομισιόν μαζί μας. Η γνώση Ζητώ συγγνώμη που δεν σας αναγνώρισα νωρίτερα, θα σας δώσω το λόγο όμω αμέσω. Λοιπόν, για να συνεχίσω από την παρατηρήση που έκανε ο κύριος De Jong. Ένας τομέας, ο οποίος ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ε, Επιτροπή μας, είναι το θέμα με τις συμφωνίες ε, διανομής, η αποκλειστική διανομής. Ποιοι είναι οι γενικοί κανόνες, ακόμα και στον τομέα των αυτοκινήτων. Θα θυμόσαστε ότι ε, όταν αναθεωρήθηκαν οι κανόνες στον τομέα των αυτοκινήτων, έπρεπε να οργανώσουμε και μια ακρόαση για να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες στους καταναλωτές. Ξέρω ότι η Κομισιό δημοσίευσε ένα κείμενο με κατευθυντήριες γραμμές για το πώς εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες, κυρίως στην, στις υπηρεσίες που παρέχονται στον τομέα της, ε, των, ε, της πόλης των αυτοκινήτων και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να σχολιάσουμε και κάποιες πτυχές του θέματος. Ε, εμείς ε, ε, είμαστε η συνείδηση του Κοινοβουλίου και έτσι πρέπει να λειτουργούμε, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει διαφάνεια. Επίσης υπάρχει και το θέμα που έθιξε και ο κύριος Ντεγιόγκ για τις σχέσεις που υπάρχουν στην αλυσίδα ε, προμήθειας ανάμεσα στους μεγάλους πελάτες, στις μικρές επιχειρήσεις και πόσο διαχειρίζονται, γίνεται διαχείριση αυτών των σχέσεων. Και ε, εδώ έχουμε κάνει δουλειά και η κυρία Κορεταμπίλη είναι υπεύθυνη για τις ε, αγορές του λιανικού εμπορίου και θα υπάρχει μια ανακοίνωση από τη Γενική Διεύθυνση για την Αγορά, για την στρατηγική στην αγορά και ξέρω ότι ο κύριος Τσόλος έχει αναμειχθεί σε θέματα που αφορούν τη διατροφική αλυσίδα. Όλα αυτά τα θέματα, επομένως, πιστεύω ότι θα προσθέσουν ε, μια κάποια αξία, ουσιαστική αξία, στην ανάλυση η οποία γίνεται σε αυτή την ετήσια έκθεση, γιατί αυτές είναι πτυχές καταναλωτών με τις οποίες, τις οποίες, ε, οι οποίες μας ενδιαφέρουν. Θέλει να προσθέσει κανείς άλλος. Εάν όχι, η κυρία Μπρούμς να σχολιάσει τα όσα ακούστηκαν μέχρι τώρα. Και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Σβάμπ για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη γιατί δεν ήμασταν εδώ όταν ξεκινήσατε. Πέρυσι ήταν διαταραγμένη χρονιά και για τις οικονομικές αγορές και για τα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν πιστεύει ότι η πολιτική ανταγωνισμού είναι ένα κομμάτι της απάντησης. Θα πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για ανάκαμψη. Και θα θέλαμε να ξέρετε ότι η έκθεση που έχετε μπροστά σας είναι Ε, σε νέα μορφή και έχει νέο περιεχόμενο, έτσι ώστε να, εξηγήσει καλύτερα τις, ε, την συνεισφορά της πολιτικής του ανταγωνισμού στην ανάκαμψη. Η νέα μορφή δείχνει, παρουσιάζει μια μη εξαντλητική ε, εκδοχή των απόψεων της Κομισιόν, η θελημένα θελήσαμε να τονίσουμε τρεις βασικές, βασικούς τομείς, ε, δημοσιονομικές υπηρεσίες, ε, τροφή και αεροπορικές υπηρεσίες, που είναι ε, πολύ επίκαιρα θέματα και κρίσιμα. Δεν θελήσαμε να εξηγήσουμε τι κάναμε πέρσι, αλλά γιατί, παρέμβαμε, γιατί παρεμβήκαμε συγγνώμη, και είναι συνέπειε συνέπειες της, συνεισφορέ, της συνεισφοράς μας στην ανάπτυξη ε, της ε, Ευρώπης και στην ευημερία των πολιτών της. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θέλουμε να ασχοληθούμε και ασχολούμεθα με, τα, με, τον, ε, με τις αποζημιώσεις. Αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο θα δοθεί με το τέλος του έτους η ιδιωτική αποζημίωση. Οι καταναλωτές ε, ε, είναι πάντα στο προσκήνιο για μας, αυτούς θέλουμε να υποστηρίξουμε και η πτυχή των καταναλωτών λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις ε, πτυχές των αποζημιώσεων και των συλλογικών αποζημιώσεων κυρίως. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του έτους έχουμε υιοθετήσει το, τα κείμενα. Μετά άκουσα και σχόλια για την εσωτερική αγορά. Η εσωτερική αγορά είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι ε, εμείς ε, ε, που ασχολούμεθα με την πολιτική ανταγωνισμού θεωρούμε ότι η ενιαία αγορά είναι ο σκοπός και ο στόχος όλων των ενεργειών μας. Επί όμως δεν έχουμε τέτοιου είδους νομοθετικές αρμοδιότητες, μόνοι μας να δρούμε. Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες που υιοθετούνται ε, σε επίπεδο ε, ε, Κομισιό. θα υπάρχει και η, η, ενιαία, η πράξη για την ενιαία αγορά υπαριθμών 2 και υπάρχουν και οι, οι εφαρμοστικές και υποστηρικτικές πράξεις. Άκουσα το σχόλιο για τις ε, σχέσεις ε, business to business. Ξέρετε ότι παρακολουθούμε πώς λειτουργούν τα κράτη-μέλη. Υπάρχει η ομάδα υψηλού επίπεδου που θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό φέτος ε, και υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών ανταγωνισμού που προσφέρουν στην Κομισιόν λεπτομέρειες για, τις, ε, ε, για την νομοθεσία που εφαρμόζουμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Και η Κομισιό θα ενημερώσει όλους για, την, για τις εξελίξεις, συγγνώμη, που είχαμε κυρίως αναφορά αφορά τις, τις τιμές των τροφίμων και όπως έχουν εξελιχθεί αυτές τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι η νέα μορφή της έκθεσης βοηθά ιδιαίτερα. Ο κύριος Σάντσιος Πεσέντιο έχει εστιάσει την προσοχή του σε κάποιες πτυχές, αλλά υπάρχουν και άλλα σημεία τα οποία θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε. Λοιπόν, κύριε Σβάμπ. Και πάλι ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε άμεσα για τη σαφήνεια των πραγμάτων. Στην έκθεσή μας μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε μόνο για αυτά τα θέματα σε αυτή την ετήσια έκθεση για τον, το δίκαιο του ανταγωνισμού που άμεσα συνδέονται με τα θέματα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Υπάρχουν πολλά βέβαια ενδιαφέροντα θέματα, αλλά για λόγους που από πλευράς κανονισμού περιοριζόμαστε δεν μπορούμε επί παντός του επιστητού να γνωμοδοτούμε. Γι' αυτό θα ήθελα να διαφωνήσω με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό που είναι η μόνη γενική ε, ε, διεύθυνση που δεν λέει μπορεί να δράσει άμεσα. Είναι η μόνη που μπορεί άμεσα να δράσει και έχει και το προτέρημα ότι η ίδια μπορεί να αποφασίσει τι θα κάνει και πώς θα δράσει. Όλα αυτά σε σχέση με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού που είναι μία από, ένας από τους πιο αποτελεσματικούς θεσμούς στην Ευρώπη για τις επιπτώσεις της ενιαίας εσωτερικής αγοράς σε ένα πολύ ευρύ πλαίσιο ρυθμιστικό και κανονιστικό, ίσως υπερβολικά ευρύ και όπως είπε ο κύριος Χατζημαρκάκης δεν καλύπτει επαρκώς το κεκτημένο και το κοινοτικό και εκτιμένο. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να εργαστούμε όχι μόνο το δίκαιο για τον ανταγωνισμό να είναι γνώμονας και μέτρο ε, στάθμισης, είναι φυσικό ότι μόνο ένα ευρύτερο πλαίσιο μπορεί να θεσπίζεται που θα εμπλέκει ιδιαίτερα την ενιαία εσωτερική αγορά. Δεύτερον, οι καταναλωτές στο δίκαιο του ανταγωνισμού διαδραματίζουν σε πολλά σημεία ένα σημαντικό ρόλο. Οι καταναλωτές γυναίκες και άνδρες και μέσα στο πλαίσιο του λιανικού εμπορίου για παράδειγμα που αναφέρθηκε από τον κύριο Ντεγιόγκ, και στις ενέργειες μεταφορές που στη σύντομη εισαγωγή μου δεν, δεν, το, δεν αναφέρθηκε και εδώ υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία αναφύονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι ιδιαίτερα όσον αφορά τη μεταφορά αγαθών με αεροπλάνα θέτει θέματα για τα ε, και εδώ υπάρχει και το αίτημα για την συγχώνευση UPS με άλλη εταιρεία. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν επιπτώσει στους καταναλωτές όταν δημιουργείται δεσπόζων ρόλος στην αγορά, κυρίαρχος ρόλος στην αγορά για κάποια επιχείρηση ή πάροχο. Κάτι πρέπει να γίνει και για τις επιδοτήσεις και ενισχύσεις εν παραλίλω ως ε, σημαντικό θέμα αυτής της έκθεσης και ταυτόχρονα και για το δίκαιο ε, το οποίο ε, εμπλέκεται εδώ. Είμαι ευγνώμων και στην κυρία Πρέντεγκαστ και στους άλλους συναδέλφους. Θα δούμε τα θέματα τα οποία συνδέουν αυτά τα θέματα στη γνωμοδότηση ώστε για την κύρια αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή έγκαιρα να είμαστε έτοιμοι για την ψήφιση. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much. So... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σβάμπ, νομίζω ότι μας υποσχεθήκατε την έκθεσή σας για μετάφραση μέχρι τέλος Οκτωβρίου. 5 ε, και 6 Νοεμβρίου θα, θα εξεταστούν εδώ. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου υποβολή τροπολογιών και μετά 17 ε, Δεκεμβρίου θα περάσει από την Ολομέλεια Επομένως, ε, περιμένουμε να, να δούμε μάλλον την έκθεσή σας ε, και ευχαριστώ και την Κομισιό που ήταν εδώ και το συζητήσαμε το θέμα. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, ήθελα να είμαι σίγουρος ότι έχουμε όλους ε, τους υπεύθυνους για την επόμενη έκθεση μαζί μας. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είναι εδώ. Θα απαντήσει στις ερωτήσεις που έχουμε για την οδηγία για την εφαρμογή της πίστοσης για τους καταναλωτές. Έχουμε υποβάλει κάποιες ε, τροπολογίες ε, εγκαίρως. Η οδηγία αυτή ήταν δική μας ευθύνη και ξεκινήσαμε από την προηγούμενη θητεία και εγώ και η κυρία Ρούλερ είχαμε εργαστεί στην αρχική πρόταση. Η έκθεση αυτή είναι μια συνεισφορά στο έργο της Κομισιόν. Η κυρία Σασόλσκα ίσως να μας δώσει μια ιδέα για το, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τι μπορούμε να περιμένουμε για την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Κόλιν Λάγκεν, την εισηγήτριά μας, να μας μιλήσει λίγο για τις τροπολογίες που υπευλήθηκαν και μετά ο κύριος Χατζη, Χατζημαρκάκης, ο οποίος θα μιλήσει για τον κύριο Μπρεζόη. Η κυρία Ρούλερ είναι εδώ. Εγώ είμαι σκιώδης για τη δική μου ομάδα και ο κύριος Ντεγιόγκ είναι σκιώδης. Λοιπόν, ας ακούσουμε καταρχάς πρώτα την κυρία Κόλιν Λάγκεν την κυρία Ντεμπέτεργκαρστα τους υπολείπους και μετά την Κομισιόν. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, όπως προαναφέρθηκε, εδώ πρόκειται για την οδηγία για τις πιστώσεις σε σχέση με τους καταναλωτές. Στις 7 Ιουνίου παρουσιάστηκε η έκθεση και ουσιαστικά δύο στόχους ακολουθεί. Ένα υψηλό επίπεδο για την προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση των διασυνοριακών συνιστοσών για τις πιστώσεις καταναλωτών. Το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών με το εναρμονιστικό πλαίσιο σε κάποια σημεία έχει αυξηθεί σημαντικά. Η διασυνορική αύξηση των πιστώσεων είναι μάλλον ασήμαντη, μόνο ένα 2% και ε, σε σχέση με το συνολικό πλαίσιο. Όλα αυτά σε σχέση με το ότι λίγες, λίγες τράπεζες προσφέρουν τέτοιου είδους δυνατότητες διασυνοριακά. Είχαμε συρρήκνωση ή μείωση λόγω της κρίσης και πολλά άλλα προβλήματα όπως η έλλειψη προσωπικών επαφών φαίνεται ότι είναι και ένα πρόσθετο εμπόδιο. Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα ήταν το πλαίσιο υλοποίησης μέσα σε μια διετή περίοδο οι διεργασίες είναι ιδιαίτερα περίπλοκες και σύνθετες και από τον εθνικό νομοθέτη και από θεσμικά όργανα πρέπει να υλοποιηθούν. Ο χρόνος πίεζε και ήταν υπερβολικά ε, σύντομος και μάλλον μια περίοδος τριετής αντί μιας διετούς περίοδου πρέπει να εισαχθεί. Εδώ επί της ουσίας αναφέρονται κάποια θέματα όπως ε, ε, η ενημέρωση, η πληροφόρηση όσον αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις των καταναλωτών. Ε, είχαν ασκηθεί επικρίσεις για υπερβολικά μεγάλο εύρος αυτής της ενημέρωσης πληροφόρησης. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ναι, έχει υποβάλει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που όμως δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Θα ήταν ευκταίο η διαδικασίες και διεργασίες αυτές να είναι για όλες τις πτυχές ταυτόσιμες σε όλες τις χώρες. Εδώ υπάρχουν προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν, για παράδειγμα σε αυτά τις προθεσμίες, πότε θα ξεκινούν και πότε θα εκπνέουν. Για αυτά τα προβλήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξέτασε τις ε, πολλές αυτές οδηγίες και διατάξεις ε, και μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι αυτή η οδηγία αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο και θεμέλιο για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρώπη. Πρόεδρε, αυτά είναι τα ουσιαστικά στοιχεία της έκθεσής μου. Για την έκθεση αυτή κατατέθηκαν 29 τροπολογίες. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχαμε μια συνάντηση σχεδόν εισηγητών σε αυτό το σημείο θα ήθελα ρητά και κατηγορηματικά να ευχαριστήσω για τον ανοιχτό και ειλικρινό δίκαιο και ε, ειλικρινή τρόπο συζήτησης ε, για αυτές τις τροπολογίες. Χαιρετίζω κάποιες πιο συγκεκριμένες προτάσεις ε, ή τοποθετήσεις τροπολογίες όσον αφορά τις πιστώσεις όσον αφορά πιστώσεις σε ξένα νομίσματα για τις δικές μου τροπολογίες είχα ήδη διατυπώσει κάποιες συμβαστικές τροπολογίες που παρουσίασα στη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών και είμαι πεισμένη ότι σε δύο-τρία περισσότερα περαιτέρω σημεία θα εξευρεθούν συμβιβασμοί. Δύο τροπολογίες δημιουργούν κάποια ερωτήματα, κάποια ερωτηματικά. Η τροπολογία 17 και η τροπολογία 21 αφορούν ερωτήματα, ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τη 17 Πιστεύω ότι ρητά θα πρέπει στο άρθρο 14 να γίνεται αναφορά και εκεί να ρυθμίζεται το περιεχόμενο αυτού, του, αυτής της πρότασης. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τοποθετηθεί από αυτού. Για την 21 κυρία Πρέντεγκάστ λέτε ότι υπάρχει πρόσθετο κόστος και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάλι θα έπρεπε να τοποθετηθεί. Κάποιες λίγες άλλες τροπολογίες δεν είναι αποδεκτές για μένα όμως όταν βλέπουμε ότι οι τροπολογίες αυτές ξεπερνούν το πλαίσιο εφαρμογής αυτής της οδηγίας και δημιουργείται η εντύπωση μιας αναθεώρησης ή μεταρρύθμισης και δημιουργούνται κάποιες ανησυχίες. Παράδειγμα, οι, ε, οι για υποθήκες στεγαστικών δανείων και έχω την άποψη ότι σε σχέση με αυτά τα θέματα η διεύρυνση για στεγαστικά δάνεια είναι ένα ουσιοδέστατο σημείο. Όμως πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να έχουμε ένα μονιμότερο χαρακτήρα αυτού του πλαισίου. Αν αληθεύει ότι λιγότερο από 2% έχουμε διασυνοριακό πλαίσιο αυτών των πιστώσεων, τότε είναι αναγκαίο όχι τώρα άμεσα να σκεφτούμε για περαιτέρω τέτοιες ρυθμίσεις που έχουμε κάποιες ρυθμίσεις σήμερα στη διάθεσή μας που πρέπει αυτές πρώτα να εφαρμοστούν προτού εισαγάγουμε νέες ε, ρυθμίσεις. Μετά μπορούμε να αφήσουμε ένα χρονικό διάστημα να ισχύσει ώστε με νυφάλιο τρόπο να εξετάσουμε το τι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό δεν πρέπει να θίξουμε ή να αλλοιώσουμε αυτή την οδηγία περαιτέρω και πρέπει να έχουμε συζήτηση με τους γεώδεις εισηγητές που είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε επί των τροπολογιών αυτών που δημιουργούν την εντύπωση αναθεώρησης αυτής της οδηγίας. Να τα ξανασυζητήσουμε τα θέματα και να δούμε αν θα βρούμε μια κοινή γραμμή πλεύσεως Συνολικά είμαι κατηγορηματικά υπέρ του να αναμείνουμε πρώτα, να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα, να δουν οι τράπεζες πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, να δουν οι καταναλωτές πώς μπορούν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους και τότε θα έχουμε την ευκαιρία να ξεπεράσουμε αυτό το όριο του 2%. Αυτή η γνωμοδότηση, Πρόεδρε, αφορά και τη γνωμοδότηση για την Επιτροπή ΕΚΟΝ το ίμιση των τροπολογιών μπορούμε να το κάνουμε δεκτό. Πάντα όμως όταν το όριο δεν δημιουργεί αναθεώρηση οδηγίας, δεν δημιουργεί εντύπωση για αναθεώρηση ή μεταρρύθμιση οδηγίας, ιδιαίτερα για τα στεγαστικά δάνεια. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Good. Well, thank you very... Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις σαφείς εξηγήσεις σας, για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε και η κυρία Πέντρεγκάστ θα πάρει το λόγο τώρα γιατί έχει υποβάλει μια σειρά πολύ ενδιαφέρουσων τροπολογιών και είχε χρόνο να ορίσει την, να, να παρουσιάσει τη θέση της. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κόλιν Λάγκεν για την εργασία της πάνω σε αυτή την έκθεση. Μετά την συνάντηση των σκιωδών ε, εισηγητών υπήρξε μια σιωπηρή συμφωνία να ε, βελτιώσουμε και να πλουστεύσουμε την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Θα ήθελα όμως να διευκρινίσω τη θέση μου για την τροπολογία 17 και να μας εξηγήσει η Κομισιόν της απόψης της, διότι υπάρχουν ανησυχίες όπου όταν ένας καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν επιπιστώσει. Αυτό δεν ε, ε, εμπίπτει στην οδηγία, διότι είναι σχέση ανάμεσα στον καταναλωτή και στο, τρα... και τραπεζικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Όμως, Πολλές φορές υπάρχουν όμως υψηλά επιτόκια, υψηλή φόρη και άλλα ποσά τα οποία ε, επιβάλλονται χωρίς να έχει υπάρξει συμφωνία. Θέλετε να σχολιάσετε και άλλα σας τροπολογίες, λέει ο πρόεδρος. Όχι, θα ακούσω πρώτα τι θα αλεχθεί και μετά νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να διευκρινίσουμε τις τροπολογίες. Αλλά και φαντάζομαι ότι όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση θα έχουμε προχωρήσει αρκετά. Ευχαριστώ πάντως πολύ που μου δίνει το, τη δυνατότητα να... Α, ο κύριος Χατζημαρκάκης έχει το λόγο. Κυρία Ρούλα. Η κυρία Ρούλα, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την... Α, όχι, εντάξει, συνεχίστε εσείς. Ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή συνεργασία και για τις προτάσεις. Για μας το θέμα αυτού του ξένου συναλλάγματος ε, είναι σημαντικό γιατί υπήρξαν προβλήματα σε κάποια κράτη-μέλη με αυτό. Και για το θέμα της ερώτησης κυρίας, ε, του θέματος της κυρίας Πρέντεγκας δεν ξέρω αν είναι μια καταχρηστική πρακτική ή αν είναι καταχρηστική εφαρμογή, ε, λαθασμένη εφαρμογή, διότι είχαμε εξαιρέσει το πεδίο εφαρμογής ε, στην ευρωπαϊκή ρύθμιση. Γι' αυτό με ενδιαφέρει άμεσα η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας πει σε τι οφείλεται αυτή η κατάσταση. Σε μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην σωστή πορεία. Θέλω να υποστηρίξω τη συνάδελφο σε αυτό που είπε. Δεν έχει ε, νόημα μετά από την μεταρρύθμιση να, ζητούμε μεταρρύθμιση οδηγιών μόλις άρχισε να εφαρμόζεται αυτή η οδηγία στα κράτη-μέλη και δεν έχουμε αρκετή πείρα σε σχέση με αυτήν. Και φυσικά για την εμβέλεια αυτής της ε, ε, πρακτικής ε, είναι περιορισμένη και δημιουργείται μεγαλύτερη σύγχυση για τους καταναλωτές και όχι βεβαιότητα και ασφάλεια αν αλλάζουμε διαρκώς τα πλαίσια. Ευχαριστώ για μια θετική έκθεση. Κύριος Χατζημαρκάκης τώρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ο κύριος Μπουσόη με παρακάλεσε να ζητήσω συγγνώμη για την απουσία του. Συμφωνεί με την δράση της εισηγήτριας ουσιαστικά. Έχει και κάποιες τροπολογίες που συνέταξε. <clears throat> Αναφέρθηκε ότι υπάρχει υποστήριξη για αυτές τον ενδιαφέρει η καλύτερη πληροφόρηση και ενημέρωση για τους ε, όσους ζητούν δάνεια και πιστώσεις ε, διασυνοριακά. Ένα ε, Consumer Information System θα μπορούσε να βελτιωθεί ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πιο ευκολότερης πρόσβασης σε τέτοιες πιστώσεις και δάνεια για αυτά που αναφέρθηκαν ότι δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια αναθεώρηση αλλά καλύτερη εφαρμογή σήμερα συμφωνώ αυτό είναι το ουσιοδέστερο ευχαριστώ να προσθέσω κάποια σχόλια δικά μου. Γιατί είμαι σκιώδη συζητητή τη ομάδα μου και κάποιο ο οποίο έχει εργαστεί πάνω σε αυτή την πρόταση από την αρχή. Η έκθεση της κυρίας Κόλλιν ε, Λάγκεν ε, αντικατοπτρίζει τις απόψεις μου επί του θέματος. Γιατί αν δείτε όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, η διασυνοριακή αγορά για την καταναλωτική πίστη δεν έχει αναπτυχθεί πάρα πολλά και γι' αυτό υπάρχουν πολλοί λόγοι, καταρχάς και για την ε, καταναλωτική εμπιστοσύνη, για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Ε, για πίστοση η οποία γίνεται, ε, σε, αναλαμβάνεται σε άλλη χώρα, σε άλλο νόμισμα. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά ρυθμίζονται από τις διατάξεις οδηγίας. Με αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα, πιστεύω ότι μέχρι στιγμής είμαστε σε πολύ αρχικά στάδια μιας ενδυνάμει αναπτυσσόμενης αγοράς ε, για το μέλλον. Και η εφαρμογή αυτής της οδηγίας φαίνεται να, να είναι λίγο άνηση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσει η Κομισιόν με τους των κρατών μελών. Υπάρχουν κάποιες αρχικές ευθύνες όσον αφορά την πίστοση για την αγορά κατοικίας ε, η Επιτροπή μας ήθελε να παρακολουθήσουμε το θέμα μέσα, τα μέσα στο πλαίσιο της οδηγίας για την κατανοητική πίστη, χωρίς όμως να μπούμε σε ξεχωριστές, σε συγκεκριμένες διαδικασίες, διότι ούτως ή άλλως διέπεται αρκετά αυστηρά η αγορά κατοικίας. Επίσης, ήθελα να πω ότι υπάρχουν κάποιες συζητήσεις για το πώς παρουσιάζεται και για το κατά πόσον παρουσιάζεται με σαφή τρόπο η πληροφορία στον καταναλωτή και κατά πόσον ο καταναλωτής την κατανοεί την πληροφορία αυτή. Επίσης, οι συνάδελφοί μου ε, έθιξαν και τα θέματα της ε, αθέμητης συμπεριφοράς ε, των οικονομικών παραγόντων στην αγορά. και υπάρχει και μια οδηγία για τις αθέμητες ε, συμπεριφορές που πρόκειται να δημοσιευθεί άμεσα και εδώ υπάρχει μια επικάλυψη. Οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές ε, καλύπτονται από συγκεκριμένη οδηγία. Ακόμα και η τιμολόγηση κάποιου προϊόντος ε, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αυξάνεται η τιμή γιατί μετά το αποσύρουν. Τέλος πάντων, η κανονική πίστη είναι ένα τομέα. που αφορά άτομα τα οποία δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ε, που καλούνται να πληρώσουν, ε, που καλούνται να δανειστούν κάποια χρήματα και να, τα, και να πληρώσουν συγκεκριμένα επιτόκια ε, εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όσον αφορά τους καρχαρίες δανειοδότες, ε, την παράνομη, ε, παράνομη δανειοδότηση και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να ρυθμίσουμε και να ελέγξουμε την παροχή δανείων σε κάποιες περιοχές. Το έχω συζητήσει το θέμα και με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, λοιπόν, ε, πρέπει οι δυνατότητες παροχής πίστοσης να χρησιμοποιούνται από καταναλωτές που είναι πολύ καλά ενημερωμένοι, που είναι πληροφορημένοι και πιστεύω ότι η ενημέρωσή τους είναι το βασικό, η βασική μας αρμοδιότητα, αλλά και το βασικό προνόμιο που έχουν αυτοί οι καταναλωτές, να είναι καλά πληροφορημένοι και ενημερωμένοι. Και θα πρέπει οι δανειοδότες να λειτουργούν με έναν σαφή και διάφανο τρόπο, με υπαλλήλου που να είναι καλά ενημερωμένοι ε, και θα πρέπει να ε, ρυθμίζονται οι δραστηριότητές τους από την ε, ρυθμιστική αρχή των κρατών μελών. Η κυρία Κόνι Λάγκεν πιστεύω ότι θα τις καλύψει όλες αυτές τις πτυχές. Και χωρίς ε, να μακρηγορήσω περισσότερο, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν να μας πει ποια είναι η θέση της Κομισιόν και μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Κόλιν Λάγκεν για να ολοκληρώσει. Αν μου επιτρέπετε πρώτα απ' όλα να συμμεριστώ μαζί σας την γενική μας εντύπωση και προσέγγιση για το πώς λειτουργεί αυτή η οδηγία στην πρακτική εφαρμογή. Τι κάνουμε τώρα και ποια θα είναι τα μελλοντικά επόμενα βήματα. Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι υπάρχει μείζον πρόβλημα με την λειτουργία, εφαρμογή και συμμόρφωση με αυτή την οδηγία. Από πλευρά της κυρία Λάγκεν αναφέρθηκε το θέμα ΣΟΥΙΠΑ ανακαλύψαμε κάποια στοιχεία τα οποία εντοπίσαμε. Τώρα θα έχουμε μια μελέτη για την αγορά και βρισκόμαστε στο μεσοδιάστημα προς ε, την ολοκλήρωσή της έχουμε συνειδητοποιήσει που έγινε τα πιο ε, ευάλωτα σημεία. Έχουμε ήδη κάνει κάποια βήματα και έχουμε κάνει κάποια διαβήματα. Αναφέρθηκε το θέμα του, ε, των εναρμονισμένων υπολογισμών για τα ποσοστά και τους, τα αριθμητικά μεγέθη. Υπήρξε μια νέα οδηγία τον Νοέμβριο πέρσι που άλλαξε το παράδειγμα ακριβώς για τους υπολογισμούς αυτούς, διότι διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν νέα προϊόντα στην αγορά που θα έπρεπε να καλύπτονται σε σχέση με αυτά που δεν καλυπτόντουσαν προηγούμενα. Τα κράτη-μέλη θα έχουν χρόνο μέχρι τα τέλη του έτους για να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν ε, την ε, οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα δούμε ποια θα είναι τα τελικά αποτελέσματα. Ήδη εφέτος το Μάιο δημοσιοποιήσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές, ε, τα στοιχεία για τον υπολογισμό αυτών των δανείων και πιστώσεων κάποια στοιχεία δηλαδή του πώς μπορούν να παρέχονται πληροφορίες και στοιχεία επ' αυτών των συνιστοσών. Είναι επικοδομητικό για τις εθνικές αρχές λοιπόν να έχουν στη διάθεσή του αυτές τις κατευθυντήρες γραμμές μέσα αυτούς τους προσανατολισμούς στη δράση τους. Επίσης έχουμε υπόψη μας για του χρόνου 2013 να αναπτύξουμε μια εκστρατεία ενημέρωσης και κατάρτισης, επιμόρφωσης, πώς όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται και να υλοποιούνται και πώς για παράδειγμα ε, μια εκστρατεία κατάτησης και εκπαίδευση θα μπορούσε σε κάποια κράτη-μέλη να δραστηριοποιηθεί, να λειτουργήσει επί των πιο ε, σημαντικών αυτών θεμάτων για τα πιο ευάλωτα αυτά θέματα. Όπως σε σχέση με το άρθρο 27 της οδηγίας θα δημοσιοποιήσουμε τη Γενική Έκθεση για την υλοποίηση και εφαρμογή αυτής της οδηγίας για τα σημεία τα οποία εξειδικεύονται σε αυτό το άρθρο, δηλαδή τα κατόφλια και τα ποσοστά κατοφλίων και το πώς θα μπορούν τα κράτη-μέλη να δρουν στη διακριτική τους ευχέρεια. Να έχουμε μια ευρύτερη εικόνα που θα απεικονίζεται για το πώς λειτουργεί η αγορά για παράδειγμα και για το ποιο θα είναι το εύρος των διασυνοριακών ε, πωλήσεων και συναλλαγών. Δεν έχουμε ε, κάποια συγκεκριμένα εξειδικευμένα στοιχεία και γι' αυτό είναι δύσκολο να εξειδικεύσει κανείς ε, ποιο είναι το πλαίσιο των διασυνοριακών τέτοιων δανείων και πιστώσεων. Οι καταναλωτές δεν συνειδητοποιούν αν οι κάποιοι πάροχοι ε, προέρχονται από κάποιες εθνικές τράπεζες. Έχουν και κάποιο τίτλο που μπορεί να είναι τίτλος αλλοδαπού κράτους ή άλλης επωνυμίας σε σχέση λοιπόν με τις αλλαγές δεν, βλέπουμε να υφίστανται λόγοι για αλλαγές. Δεν προτιθέμεθα να ε, προτείνουμε αλλαγές ε, σε σχέση με την οδηγία. Είναι πολύ πρόημο να γίνει κάτι τέτοιο. Ακόμα ένας ενάμισης χρόνος έχει περάσει, ούτε καν δύο χρόνια. Είναι δύσκολο λοιπόν μέσα σε ένα τέτοιο διάστημα να δει κανεί ε, προς ποια κατεύθυνση πρέπει να, κάτι να αλλάξει ή όχι. Έχουμε και κάποια συγκεκριμένα εξειδικευμένα ερωτήματα από τους ευρωβουλευτές ε, που διατυπώθηκαν και θα ήθελα να απαντήσω σε αυτά. Το πρώτο, η πρώτη παρέμβαση για την τροπολογία 17. Για αυτή την τροπολογία αυτή η τροπολογία αφορά τα κόστη σε σχέση με την ε, υπαναχώρηση όσον αφορά μια συμφωνία ε, δανειοδότησης. Σαφώς αναφέρεται στο άρθρο 14 14-3 εδάφιο 3 της οδηγίας, ότι μόνο και αποκλειστικά αιτήματα των ε, πιστωτών σε σχέση με τέτοιου είδους δάνεια μπορούν να καλύπτονται μέχρι τη στιγμή υπαναχώρησης. Οποιεσδήποτε άλλες ε, πληρωμές, ε, για παράδειγμα τέλη, προμήθειες ε, κτλ. δεν μπορούν να επιστρέφονται. Εκείνα τα οποία μπορούν να επιστρέφονται είναι σε σχέση με τα τέλη έναντι των δημοσίων αρχών οποιαδήποτε άλλα τέλη θα πρέπει να επιστρέφονται στους ε, καταναλωτές. Και επιπλέον σε σχέση με την αιτιολογική σκέψη 34 αναφέρεται ότι η παναχώρηση θα πρέπει να είναι χωρίς κύρωση, χωρίς ε, ποινή εις βάρος ε, του δανειζομένου. Με βάση αυτά τα στοιχεία νομίζω ότι απαντούμε στο ερώτημα που διατυπώθηκε. Υπήρξε επίσης και το ερώτημα για καλύτερη, το ζήτημα για καλύτερη πληροφόρηση σε περίπτωση διασυνοριακών δανείων και πιστώσεων, ιδιαίτερα για την καλύτερη κατανόηση από πλευράς των δανειστών τι θα συνέβαινε σε σχέση με δάνεια σε ξένο συνάλλαγμα και σε σχέση με τις, ε, ε, ε, τους όρους αλλοδαπής όσον αφορά τα επιτόκια. Αυτά είναι τα ε, πληροφοριακά στοιχεία που αποτελούν επεξηγήσεις μάλλον προς κατανόηση, προς καλύτερη κατανόηση ε, για τους καταναλωτές. Ο κίνδυνος δεν μπορεί να καλύπτεται με αυτόν τον τρόπο κατά 100% υφίσταται κίνδυνος. Τώρα, αν θα, ε, πράγματι θα επισυμβεί αυτό ή όχι, είναι κάτι διαφορετικό. Επαρκείς επεξηγήσεις πρέπει να, να δίνονται για το τι μπορεί να επισυμβεί σε διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά αυτές τις, ε, αυτούς τους όρους ε, δανείου σε ξένο συνάλλαγμα. Δεν είμαι βέβαια να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις και παρεμβάσεις και σχόλια. Αυτά είχα υπόψη να πω, αυτά έχω σημειώσει ε, στις σημειώσεις μου και αυτά είχα να σας πω. Έχει κάποιος κάποιες άλλες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρεί κάποιος ότι κάτι δεν απαντήθηκε. Όλοι είναι ικανοποιημένοι από ό,τι φαίνεται. Έχετε κάτι για να ολοκληρώσετε για το χρονοδιάγραμμα. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες επισημάνσεις για τη μελέτη σας. Πότε θα υπάρξουν κάποιες ε, αλλαγές, ε, κάποια ε, μεταρρύθμιση είμαστε υποχρεωμένοι να δημοσιοποιήσουμε αυτή την έκθεση που θα καλύπτει τα στοιχεία αυτής, ε, τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης και του ελέγχου εφαρμογής ε, όσον αφορά την ε, συμμόρφωση και υλοποίηση αυτής της οδηγίας στα κράτη-μέλη μέχρι το Μάιο 2013, όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 27 της οδηγίας. Και φυσικά θα προετοιμάσουμε και τις ε, εσωτερικές μας μελέτες όπως απαιτείται για αυτό το πλαίσιο αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Ήταν μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Εσείς κύριε Κόρμεν Λάγκεν θα θέλατε να ολοκληρώσετε από πλευρά σας. Μπορώ και πάλι πολύ σύντομα να αναφερθώ σε αυτά. Χαίρομαι για το όσα μας εξήγησε η προλαλή σας για την τροπολογία 17 διότι και εγώ το άρθρο 14 εδάφιο 3 έτσι το διάβασα και το ερμήνευσα, διότι αυτά τα οποία σίγουρα για τη Μεγάλη Βρετανία ε, αναφέρονται δεν ανταποκρίνονται απόλυτα με αυτή, σε αυτή την οδηγία. Τώρα έχουν αποσαφινιστεί περισσότερο αυτά τα πράγματα και για το σύστημα ενημέρωσης πληροφόρησης γίνεται δεκτή τροπολογία Μπουζόη και έτσι νομίζω με τις περαιτέρω συζητήσεις που θα έχουμε κυρία Πρένταγκάστα θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε ένα συνενετικό πλαίσιο για αυτή την οδηγία, για αυτή την έκθεση και να ψηφίσουμε συνενετικά. Ευχαριστώ. Sorry, I'll put the microphone We're going to vote. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή 11 Οκτωβρίου και θα, ε, στις 10 Οκτωβρίου θα εξετάσουμε τις ε, τροπολογίες και θα έχουμε μια έκθεση... Α, έχουμε τη γνωμοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής. Ωραία. Έχουμε την έκθεση από την Οικονομική Επιτροπή την οποία πρέπει να εξετάσουμε και μετά θα... ο στόχος μας είναι να περάσει από την Ολομέλεια το Νοέμβριο. Επομένω, έχουμε ε, καιρό, αν θέλετε, να πιέσουμε την Κομισιό να συνεισφέρει περαιτέρω και να μας δώσει μια περαιτέρω γνωμοδότηση όταν μας στείλουν την έκθεση για την αναθεώρηση. Ίσως και μια τροποποιημένη οδηγία για το 2013 κάποια στιγμή. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας για σήμερα το βράδυ. Θα τα πούμε αύριο στις 9 ακριβώς για την ε, ε, εξέταση της, ε, των τροπολογιών για τις κρατικές προμήθειες και έχουμε και μία, έχουμε και μία σειρά ακροάσεων Από τις 10.30 έως τις 12 θα εξετάσουμε την οδηγία σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών. Η κυρία Βανίλε θα παρουσιάσει το απόγευμα την έκθεσή της ε, για, τις, ε, για τα επαγγελματικά προσόντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα συνεδρίασης.